<laughs> Peut-être si la présence Θα ξεκινήσουμε. Και θα μιλήσω πορτογαλικά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους, όλες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Σήμερα το πρωί έγινε μια ακρόαση, δημόσια κροάση, που δυστυχώς δεν μπορέσαμε όλοι να συμμετάσχουμε, διότι υπήρχαν και άλλες συνεδριάσεις άλλων επιτροπών, όπου διεξήχθησαν ψηφοφορίες, όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία συμμετέχω και εγώ και δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα ούτε εγώ στην ακρόαση όσον αφορά την κοινωνική κατάσταση των γυναικών στις μειονοτικές εθνοτικές ομάδες. Πρώτο σημείο έχουμε έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν προτάσεις τροποποίησεων, υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν κάποιε κάποιες παρατηρήσεις, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Δεν υπάρχει ανακοίνωση της Προέδρου, οπότε πάμε στο σημείο 3 κατευθείαν. Έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως της 28 Ιανουαρίου. Ε, τα πρακτικά έχουν διανεμηθεί. Έχετε χρόνο μέχρι το τέλος συνεδριάσεως για να υποβάλλετε αντιρρήσεις διαφορετικά θα θηρηθούν ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Επόμενο σημείο. Είναι μια σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση πρόταση της κυρίας Λούλινγκ για την ισότιμη αντιμετώπιση ανδρών γυναικών που ασκούν αυτόνομη δραστηριότητα. Όπως σημειώνεται, Η πρώτη ανάγνωση έγινε στις 6 Μαΐου του 2009 και στις 8 Μαρτίου του 2010 υιοθετήθηκε θέση του Συμβουλίου και υπευλήθη 24 Μαρτίου αυτή η θέση στο Κοινοβούλιο, κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο. Έγιναν κάποιες τροποποίησεις στην πρώτη ανάγνωση, τροπολογίες που υπέβαλε και πρότεινε το Κοινοβούλιο που υιοθετήθηκαν εν μέρη ή στο σύνολό τους από το Συμβούλιο. Πάνω σε αυτό θα ακούσουμε την κυρία Λούλινγκ, την εισηγήτρια που θα μας ενημερώσει. Έχετε το λόγο κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως σωστά υπενθυμίσατε, το Συμβούλιο χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για να μας διαβιβάσει την ε, κοινή του θέση. Δηλαδή γνωρίζαμε όμως από το τέλος Νοεμβρίου πως τα πού πήγαιναν τα πράγματα, αλλά με όλες τις ε, διαδικασίες που ακολουθήθηκαν δεν λάβαμε γνώση επισήμω της κοινή θέσεως παρά μόνο στις 8 Μαρτίου και γι' αυτό μεριμνήσαμε να σας παρουσιάσουμε τώρα ένα σχέδιο συστάσεως για τη δεύτερη ανάγνωση. Εν τω μεταξύ, συμμετείχα σε πολλές συναντήσεις με την Προεδρία, την Ισπανική, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινώς για την άριστη συνεργασία μας εν ώψη της ε, παρουσιάσεως αυτής της συστάσεως για δεύτερη ανάγνωση. Σε αυτό το πλαίσιο, από κοινού πολλές φορές διεξήχθησαν συνεδριάσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορώ να σας πω ότι προφανώς είμαστε ικανοποιημένοι για όλες τις θετικές απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά την πρότασή μας. Απομένουν όμως κάποια σημεία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως το Συμβούλιο δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τη δική μας γραμμή. Η Ισπανική Προεδρία μου εξήγησε πάρα πολύ καλά που βρίσκονται τα όρια για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποια σημεία επί των οποίων δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο λιγμών με το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να τεκμηριώσουμε τη θέση μας. Το Συμβούλιο, κυρίως όσον αφορά την προστασία, την κοινωνική των συζύγων και των συντρόφων ζωής, που θέλαμε αυτό να προβλέπεται ως υποχρέωση, και όχι προστασία κατόπιν ετήματος, ουδέμια ευελιξία εκεί, Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ασφάλιση υποχρεωτικά. Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο ελίγωμων για την επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο μέσω των δικών μας φαντάσεων. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όσον αφορά αυτή την κοινωνική προστασία στην κοινή θέση του Συμβουλίου Σημειώθηκε πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο εν συγκρίση με τα ισχύοντα τώρα, διότι το Συμβούλιο συμφωνεί να αναφέρουμε ότι όταν σε ένα κάτω μέλος υπάρχει σύστημα προστασίας, κοινωνικής προστασίας για τους ανεξάρτητους εργαζομένους, για τους αυτοτελείς εργαζομένους, ε, όταν υπάρχει ένα σύστημα όπως τα περισσότερα κράτη-μέλη, τον λόγο κάτω μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ούτω ώστε και οι σύζυγοι και οι σύντροφοι ε, να μπορούν να ωφεληθούν από μια κοινωνική προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το είχαμε στις περισσότερες χώρες μέλη. Το Συμβούλιο λοιπόν προτείνει να πούμε ότι τα κράτη-μέλη δύνανται να αποφασίσουν κατά πόσο αυτή η κοινωνική προστασία ε, εφαρμόζεται υποχρεωτικός ή εθελοντικός. Και κατά συνέπεια μπορεί να προβλέπει αυτή η κοινωνική προστασία να μην χορηγείται παρά μόνο κατόπιν αιτήματος των συζύγων ή των συντρόφων. Η μεγάλη πρόδοση είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει πρέπει να προτείνουν ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό, προαιρετικό και αν αποφασιστεί αυτό να είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό, εκείνοι που θέλουν να το εκμεταλλευτούν θα πρέπει να εμφανιστούν και να το ζητήσουν. Για τους μισθωτούς είναι διαφορετικό. Είναι ο εργοδότης ο οποίος λέει έχω ένα μισθωτό θα ασφαλιστεί. Οι αυτοτελείς επαγγελματίες, οι αυτοαποσχολούμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν. Είναι κάτι που εξυπακούεται. Συμφωνώ. Εγώ, διότι διαφορετικά δεν θα πετύχουμε κανένα αποτέλεσμα. Συμφωνώ να κάνουμε αυτό το βήμα Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στη χώρα μου, πριν την υποχρεωτική ασφάλιση, Το είχαμε αυτό στην ε, υποχρεωτικό στη Γεωργία, αλλά πριν να εφαρμοστεί αυτό και σε άλλους τομείς, βιοτεχνία, εμπόριο, ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, κάθε είδους, περάσαμε και εμείς μια περίοδο όπου μπορούσε κανείς εκουσίως ή να ασφαλιστεί ή να μην ασφαλιστεί. Οπότε, με αυτό το κείμενο του Συμβουλίου, φτάνουμε σε αυτό το στάδιο. Σημαντικό. Ακόμα και αν εγώ θα ήθελα να το πηδήξουμε αυτό το στάδιο, προχωρήσουμε πιο κάτω. Στο Συμβούλιο όμως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ελίγμων για να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό σας ζητώ να υποστηρίξετε το άρθρο 7 του Συμβουλίου και να ακολουθήσουν ιδέουσες αιτιολογικές σκέψεις. Και ένα άλλο επίτευγμα, ένα άλλο σημείο που κολλάμε μάλλον, είναι η προστασία της μητρότητας. Και εκεί το Συμβούλιο μας ακολούθησε στη θέση μας, δηλαδή ότι θα πρέπει να παράσχεται μια προστασία της μητρότητας, αλλά προφανώς δεν μπορεί να είναι η ίδια προσέγγιση όπως για τους μισθωτούς. Γι' αυτό έχει τη θέση του το κείμενο εδώ και όχι σε μια οδηγία που αφορά τους μισθωτούς. Υπάρχουν όπως λέει το κείμενο, τα κράτη-μέλη μάλλον λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, τόσο ώστε οι γυναίκες που ασκούν μία ανεξάρτητη δραστηριότητα, δεν μιλάμε μόνο για συζύγους, ανεξάρτητες γυναίκες και συζύγους ή συντρόφους των ανεξαρτήτων ούτως ώστε να μπορούν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να έχουν δικαίωμα σε ένα επίδομα, το ενδεδειγμένο επίδομα μητρότητα που θα τους επιτρέπει να διακόπτουν τη δραστηριότητά τους στην επαγγελματική για λόγους εγκυμοσύνης ή μητρότητα. Το Συμβούλιο είχε προτείνει 14 εβδομάδες, διότι ήθελε να βάλει αριθμητικό στοιχείο το Συμβούλιο και ήθελε να εμπνευστεί από τα εφιστάμενα για τους μισθωτούς. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν θέλουν αναφορά στην οδηγία για τους μισθωτούς. Θα πρέπει να βρεθεί μια διατύπωση που να επιτυγχάνει τα αποτελέσματα η οποία όμως αναβάνει υπόψη τις ευαισθησίες κάποιων κρατών που δεν θέλουν αναφορά της οδηγίας του 92. Και πιστεύω ότι μπορώ να σας προτείνω μια τροπολογία επιπλέον που θα έλεγε αγγλιστή λίγο πολύ τα εξής. Η διάρκεια της περίοδου κατά τη διάρκεια την οποία οι γυναίκες αυταπασχολούμενες εργαζόμενες και οι γυναίκες σύζυγοι σύντροφοι λαμβάνουν επίδομα μητρότητας ισοδυναμή με τη διάρκεια άδεια μητρότητας που χορηγείται στους μισθωτούς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν λέμε 14, αν πούμε 14 εβδομάδες όπως λέει η οδηγία, ή να πούμε ότι προσωμιώνεται η διάρκεια αυτή με τη διάρκεια της άδεια μητρότητας για μισθωτούς, όπως ισχύει τώρα, το ίδιο, η μία, η μία ή η άλλη. Το ίδιο πράγμα είναι. Αν αυτό παρηγορεί όμως τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν ε, ρητή αναφορά της οδηγίας, αυτό δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το δικαίωμα καλύψεως των 14 εβδομάδων. Θα προσθέταμε, θα έλεγα, εφόσον η οδηγία συζητείται ακόμα με τους μισθωτούς, σε περίπτωση, θα προσθέσαμε, που η διάρκεια της μητρότητας, της άδειας μητρότητας που προβλέπεται για μισθωτούς τροποποιηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογώντα κατά πόση η διάρκεια των επιδομάτων μητρότητα για τι γυναίκε αυταπασχολούμενε και γυναίκε συζύγου θα πρέπει και ε, αυτή να τροποποιηθεί. Ξέρουμε λοιπόν ότι αν αλλάξει η οδηγία, αν τροποποιηθεί η οδηγία περί μισθωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποχρεώσει να μας υποβάλει πρόταση που θα προσάρμοζε δεόντως το καθεστώς για τους αυταποσχολούμενους, ανεξάρτητους εργαζομένους και τους συντρόφους τους. Ελπίζω ότι με αυτό θα μπορέσουν να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη. Εγώ έκανα κάποιες αλλαγές και ξέρω ότι συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Προφανώς δέχονται τη δική μας πρόταση. Δηλαδή αυτή η οδηγία δεν αφορά μόνο τη γεωργία. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει κάτι τέτοιο, διότι δεν δημιουργεί προβλήματα λοιπόν. Η τροπολογία μας υπαριθμών ένα λέει ότι α, τροποποιούμε την οδηγία για να ενισχύσουμε την προστασία της μητρότητας των ανεξαρτήτων εργαζομένων και για να βελτιώσουμε την κατάσταση των συζύγων των ανεξαρτήτων εργαζομένων. Σαφές το κείμενο, πολύ πιο δέτερο, που θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, που λέει ακριβώς αυτό που επιθυμούμε. Επίσης, το Συμβούλιο συμφωνεί να δεχθεί την τοπολογία μας, όπου αναφερόμασταν στην, στο ψήφισμα του 97 για την ε, κατάσταση των συμβουλισσών ε, συζύγων. Απλά επαναλαμβάνουμε τις προτάσεις του 97. Τώρα η τροπολογία 3 δική μου. Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Ε, κάποια κράτη-μέλη δεν δέχτηκαν ή δεν κατάλαβαν ότι δεν θέλουμε το κείμενο του Συμβουλίου που λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν εθνικές διατάξεις που θα περιορίσουν την πρόσβαση σε ειδικά καθεστώτα προστασ... κοινωνικής προστασίας ή σε κάποιο επίπεδο προστασίας. Αυτό είναι ένα τέχνασμα, όχι τέχνασμα δηλαδή, αλλά ε, ε είναι μια ανησυχία των Γερμανών οι Γερμανοί έχουν κάποια ειδικά καθεστώτα, έτσι, πολύ ειδικά για κάποιες κατηγορίες ανεξαρτήτων ε, εργαζομένων, γιατρών νομίζω, δεν είναι υποχρεωμένοι να τα αλλάξουν. Δεν θέλουμε όμως ωστόσο να αναφέρεται αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να φύγει αυτό από την πρόταση του Συμβουλίου λιτοπολογία 4. Και εδώ ελπίζω ότι θα συμφωνήσει το Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχε προτείνει να προσθέσουμε μία φράση στο κείμενό μας επιπλέον η οικονομική κατάσταση του ατόμου ή της οικογένειας υπό εξέταση μπορεί να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό των εισφορών και των παροχών για την ένταξη στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει μεταξύ των μισθωτών και, και μισθωτοί υπάρχουν. Όχι εκατομμύρια, αλλά εγώ ξέρω μισθωτούς που είναι πολύ πλουσιότεροι από ορισμένους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Κανείς ωστόσο δεν θα τολμούσε να πει στο ΊΚΑ ότι λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική τους κατάσταση ή την περιουσία που έχουν για να ρυθμίσουμε το πώς θα μετάσχουν στην κοινωνική ασφάλιση ή όχι. Εφόσον δεν υπάρχει κάτι για τους μισθωτούς, δεν πρέπει να υπάρχει και για τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Σας είπα ήδη για την τοπολογία 5, εδώ θα κάνω μία πρόταση για να διαγραφεί η μνήμα στην οδηγία του 92 που αφορά τη μνήμα της οδηγίας δηλαδή αυτής αλλά το υπόλοιπο θα είναι ίδιο. Επί της ουσίας θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Εγώ τουλάχιστον μπορούσα να συμφωνήσω στην τροπολογία 6. Και εδώ ελπίζω να πείσουμε το Συμβούλιο να δεχθεί την τροπολογία μου. Γιατί το Συμβούλιο θέλει να πει ότι σε ό,τι αφορά την προστασία της μητρότητας, ότι οι αυτοπασχολούμενοι και οι σύζυγοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο μέτρο του δυνατού σε εγώ διαγράφω αυτή τη φράση στο μέτρο του δυνατού. Λέω ότι πρέπει να, υπά, να δίδεται πρόσβαση σε κάθε υφιστάμενη υπηρεσία παροχής προσωρινής εγκατάστασης που υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό είναι δυνατό ή όχι στα κράτη-μέλη. Εγώ ήθελα να μπει το κείμενο αυτό, γι' αυτό προτείνω την τροπολογία 6. Επίσης, πρότεινα και την τροπολογία 7 το, το Συμβούλιο μας είχε πετάξει στα μούτρα ένα κείμενο λέγοντας ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ε, προστασίας. Εγώ το ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα βιωσιμότητας, μακροχρόπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας όλων των κοινωνικών συστημάτων και των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών. Γιατί όμως να μπει σε μια οδηγία μια τέτοια φράση. Εγώ είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να πείσουμε το Συμβούλιο να διαγράψει την αιτιολογική αυτή σκέψη. Η τροπολογία 8 αφορά τους οργανισμούς. Είπαμε ότι το Συμβούλιο θέλει να υπάρχουν πάντα οργανισμοί που προσπίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εγώ το θεωρώ σημαντικό. Εγώ έχω την άποψη ότι οι οργανισμοί πρέπει να είναι ίδιοι και για τους ε, αυτοπασχολούμενους και για τους μισθωτούς. που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Τέτοι, τέτοιοι φορείς υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αν σε ένα κράτος υπάρχει ένας οργανισμός για τα κοινωνικά δικαιώματα και την προστασία της αρχής της ισότητας της μισθολογικής ισότητα. Προφανώ είναι αρμόδιος αυτός ο οργανισμός, αυτός ο φορέα, αλλά δεν θέλουμε κάτι τέτοιο στο κείμενο. Η τροπολογία 9. Δεν είμαι πεπισμένη εδώ ότι θα διδεχθεί το Συμβούλιο. Αφορά το θέμα του κατά πόσο τα κράτη-μέλη Πρέπει να συμφωνήσουμε. Πρέπει να συμφωνήσουν. Προφανώς αν θέλουμε να υπάρξει μια ε, πρόοδος, θα πρέπει τα κρατημένα να μπορούν να αποφασίσουν ότι η κοινωνική προστασία ε, εφαρμόζεται σε υποχρεωτική σε προαιρετική βάση. Εδώ υπάρχει συμφωνία. Αυτό όμω σαν συνέπεια θα έχει ότι η προστασία αυτή χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήματος του συζύγου ή του συντρόφου. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι σαφές ότι εγώ μπορεί να θέλω τη σύνταξή μου και να έχω δικαίωμα σε ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας πρέπει να υποβάλω μια αίτηση. Αλλά νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε σε συμφωνία. Να υπάρχει συμφωνία δηλαδή. Τροπολογία 10. Το ίδιο πρόβλημα είναι. Το Συμβούλιο λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσο το επίδομα μητρότητας χορηγείται υποχρεωτικά ή σε προαιρετική βάση, αλλά όπως και για την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να προτείνω είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά ένα επίδομα ε, το Συμβούλιο όμω θέλει να προσθέσει ότι αντίστοιχα μπορεί να προ... πρέπει να μπορούν να προβλέπουν ότι το επίδομα αυτό χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήματο μια γυναίκα που ασκεί ε, δραστηριότητα αυτό απασχολούμενο εργαζόμενου ε, ή είναι σύζυγος ε, ενός αυτοαπασχολούμενου ή σύντροφος. Εμένα μου φαίνεται αυτονόητο Άλλο υπάλληλο. Ο υπάλληλο λέει είμαι έγκυο, ε, παίρνω το επίδομα. Ανεξάρτητο πρέπει να το πει κάπου, δηλαδή πρέπει να πάει να το πει. Αν αρχίσουμε και γράφουμε σε όλα τα κείμενα τι είναι το σύνηθε. ή αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να το δηλώσουν. Ο υπεύθυνο οργανισμός για την αποζημίωση της μητρότητας δεν μπορεί να μυρίσει τα νύχια του ότι η κυρία Τάδε είναι έγκυος. Άρα πρέπει να το εκδηλώσει. Να πει είμαι έγκυος, θέλω το επίδομα. Τέλο αν αυτό καθησυχάζει το Συμβούλιο, δεν είμαι αντίθετη, αλλά ε, ε, πρέπει αυτό που είναι σημαντικό είναι να προχωρήσουν και να προτείνουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά μία μορφή προστασία τη μητρότητα. 11. Δεν έγινε κατανοητή νομίζω, κατανοητό το κείμενο, διότι ίσως είναι αυτό που αφορά τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε το κείμενο. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στο β και να κρατήσουμε το γ για το 8-3. Πρέπει να διευκρινίσουμε το κείμενο λέγοντας τι ακριβώς θέλουμε. Επί της ουσίας όμως δεν υπάρχουν προβλήματα. Η 12 είναι συνέπεια της αιτιολογικής σκέψης. Θέλουμε και αυτό και εδώ να φύγει το κατά το δυνατό. Το 13 είναι το αντίστοιχο των αρμόδιων φορέων και η 14 προτείνουμε η έκθεση αυτή να λαμβάνει υπόψη κάθε αλλαγή της νομοθεσίας στην Ένωση για τους μισθωτούς. Νομίζω ότι και εδώ μπορώ να προτείνω, μάλλον να σας ε, προεξοφλήσω ότι θα συμφωνήσει το Συμβούλιο. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι μπορεί να μην πετύχαμε τα πάντα, πετύχαμε ωστόσο να κουνηθεί, να μετακινηθεί το Συμβούλιο με να μετακινηθεί αρκετά. Όχι 100% προς την κατεύθυνσή μας, αλλά δεδομένων των επιφυλάξεων που υπήρχαν στο Συμβούλιο, που φάγαν ένα χρόνο να συμφωνήσουν, πρέπει να σας πω ότι αν μπορέσουμε να κάνουμε δεχτές τις τροπολογίες, θα μπορέσουμε να ελπίζουμε να περάσει η σύσταση το Μάιο για να μπορέσει η Ισπανική Προεδρία να εγκρίνει το κείμενο επί του οποίου συμφωνήσαμε πριν λήξει η Προεδρία. Άρα μπορεί να μας ε, χρειάστηκε από το 86 μέχρι τώρα να αλλάξει η οδηγία του 86 που ήταν αρκετά άτολμη. Το κείμενο τώρα είναι σημαντικό, έχει σημαντικές αλλαγές, περιλαμβάνει μεγάλη πρόοδο για τους ανεξάρτητους, ιδιαίτερα δε για τους συμβοηθούντες συζύγους και συντρόφους. Τα κράτη τώρα πρέπει να προτείνουν στην σύζυγο και στον, στη σύντροφο συστήματα. Κάτι που σε πολλά κρατημέλη δεν υφίστατο μέχρι τώρα. Ελπίζω να συμφωνήσουμε γρήγορα για τις τροπολογίες αυτές. Θα συνεχίσω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ώστε να τους πείσω για τις τροπολογίες που θέλουμε να προτείνουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Λούλινγκ για την παρουσίασή σας και πλήρη και σαφής που δημιούργησε ήδη πολλά αιτήματα ανάληψης λόγου. Η κυρία Κλάση έχει το λόγο. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ευχαριστώ. Θα πω στην κυρία Λουλίνγκ πως δεν χρειάζεται να καταθέσει 100 τροπολογίες γιατί πρέπει να μπορέσουμε και να το συζητήσουμε αλλά λέει πως υπάρχει πρόοδος και χαιρόμαστε βεβαίως για την προστασία των μητέρων οπωσδήποτε συμφωνούμε, αλλά όταν μιλάμε εδώ πέρα για κοινωνική προστασία και προστασία των ελευθέρων επαγγελματιών είναι και ένα ζήτημα αρχής. Όταν διαβάζουμε εδώ πέρα τον στόχο των τροπολογιών, τότε δεν ξέρω, δεν μπορεί εδώ πέρα να ορίζουμε ελάχιστη κοινωνική ασφάλεια και να την ορίζουμε αυτή χρηματικά στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Θα πρέπει να ζητάμε την ελάχιστη προστασία των κρατών μελών και η χρηματοδότηση να μην γίνεται μόνο από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Το να μετρήσουμε βεβαίως το εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από κάποιον ο οποίος παίρνει μισθό. Πρέπει να γίνει μια διάκριση ειδικά όσον αφορά την προστασία της μητρότητας που είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και θυμόμαστε πως ε, στο πρόσφατο παρελθόν το θέμα της ισότητας τίθεται εξή γιατί να πληρώνουν περισσότερο οι γυναίκες από ότι οι άντρες για την ασφάλιση υγείας γιατί λέγανε πως οι γυναίκες ε, αρρωσταίνουν πιο συχνά ε, ή θένε περισσότερες παροχές γιατί υπάρχει η προστασία της ε, μητρότητας. Λύθηκαν ε, αυτά τα ζητήματα όμως και πέρασαν σε μια γενικότερη ασφάλιση. Είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να φροντίζει το κράτος. Και ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Λουλίνγκ για τον τρόπο με τον οποίο τα αναφέρει και τα καταγράφει. Ε, μέχρι ενό σημείου δηλαδή πρέπει να φτάνουν οι τροπολογίε. Δεν μπορεί να λέμε πως κάποιο έχει δικαίωμα σε κάτι και... Τέλος, δεν μπορεί το κράτος να εξακριβώνει τα πάντα ή να, να ψάχνει να μυρίζει τα νύχια του πραγματικά. Νομίζω εξάλλου πως υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες οι οποίες πηγαίνουν πολύ μακριά από την κοινή θέση στις ε, διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μία εντολή στην εισηγήτρια για να μπορέσει να διαπραγματευτεί για να έχουμε μια πολύ καλύτερη διαπραγματευτική βάση και καλό θα ήταν ε, η Ισπανική Προεδρία να το ολοκληρώσει αυτό. Η κυρία Λούλινγκ ανέφερε το 1986. Το 1986 εγώ να ε, Γέννησα το τρίτο μου παιδί και εγώ είμαι. Είμαι αγρότησα, ελεύθερη επαγγελματία. Και στα δύο πρώτα παιδιά δεν έλαβα λοιπόν τίποτα. Ένα επίδομα μητρότητα στο τρίτο παιδί έλαβα μας ωφέλισε πάρα πολύ ε, μια αγροτική οικογένεια. Και αν γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Και έτσι ως μητέρα και εγώ μεγάλη πια θα χαρώ πάρα πολύ για τις νέες γυναίκες και την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλάς. Πολύτιμη αυτή η συνεισφορά που βασίστηκε στην εμπειρία σας. Η κυρία Τόμψον έχει το λόγο. Well, I would ask the floor. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο για να ε, μιλήσω εξ ονόματος κυρίας πλάμη η οποία απουσιάζει, έχει ανηλυμένη υποχρέωση στη Βιέννη. Οπότε θα ήθελα εγώ να κάνω την παρέμβαση που θα έκανε εκείνη. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή δεν υπάρχει λόγο να μειωθεί το πεδίο εφαρμογή μόνο σε αυτοαπασχολούμενε γυναίκε ή συζύγους ή συντρόφου στον αγροτικό τομέα και οι επαγγελματίε και το εμπόριο δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν επειδή επέλεξαν να δουλέψουν σε έναν άλλο τομέα και όχι στη Γεωργία, εδώ πέρα νομίζω συμφωνούμε με την κυρία Λούλινγκ. Δεύτερον, η σύνδεση των ε, γυναικών και η σχέση τους με το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Η θέση μας είναι ίδια, αλλά διαφέρει η αιτιολόγηση, καθώς το σύστημα καλύπτει την αρρώστια, την αναπηρία και άλλες περιπτώσεις βεβαίως και βεβαίω σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει φόβος για πάρα πολλά μεγάλα έξοδα. Οπότε θα πρέπει η συνεισφορά αυτή να εκπίπτει από την εφορία. Όσον αφορά, όσον αφορά την τροπολογία 3 για την βελτίωση της υγείας ε, και της ασφάλειας ε, εγγύων αυτοαπασχολούμενων. Οι αυτοαπασχολούμενες που αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί έχουν δύο μεγάλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα η απουσία τους από την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά το οποίο βέβαιω έχει άμεσο αντίκτυπο και δεύτερον το ότι δεν μπορούν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους στην περίοδο πριν και μετά. Και βεβαίως η πλειοψηφία τους εργάζονται ε, μόνος τους, οπότε δεν υπάρχει κάποιος εργοδότης για να τους κρατήσει τη θέση εργασίας, οπότε μπορούν μόνο να εξοικονομήσουν χρήματα πριν την ε, εγκυμοσύνη, κατά το οποίο είναι δύσκολο βεβαίως γιατί δεν πληρώνονται πάρα πολύ καλά, ή να συνεχίσουν να δουλεύουν μέχρι τη γέννα και αμέσως μετά. Οπότε εγώ θεωρώ πως οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να υποφελούνται του συστήματος ε, κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζεται στην οδηγία 92 ε, και επίσης ε, στην οδηγία που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων εγγύων και εδώ πέρα άκουσα την κυρία Λούλινγκ που είπε πως θα προτιμούσε κανόνες παρόμοιους με τους κανόνες της ε, Ένωσης. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται μετά με τις ε, έξι εβδομάδες ε, της υποχρεωτικής περίοδου. θα αφορά αυτό και τους αυτοαπασχολούμενους. Τέλος. Ένα φορέα που θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή. Οι διατάξει για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών θα πρέπει να αποσυνδεθούν από αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε ο φορέα, ο αρμόδιος για την εφαρμογή των διατάξεων πρέπει να είναι αυτός που έχει ευθύνη και σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης ε, μεταχείρισης και όχι ο φορέας που είναι υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε βρισκόμαστε σε μια φάση της συζήτησης σημαντική. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Λούλινγκ, διότι κατά τη διάρκεια των ετών πολλές φορές έθεσε το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις προηγούμενες ε, θητείες την είχα γνωρίσει και προεδρεύουσα της Επιτροπής είχε αναλάβει το θέμα αυτό είναι ένα πρόβλημα που 20 χρόνια συζητείται. Συνέχισε να ασκεί πίεση, ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, για ένα σημαντικό θέμα που θέλω να υπογρανίσω. Δεύτερον, συμφωνώ με την κυρία Λούνινγκ σε πολλά θέματα. Όταν αναφέρει ότι πρέπει να αφορά όλους τους αναφέρει να αφορά η ρύθμιση αυτή όλες τις ε, γυναίκες ε, που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα και όχι μόνο στη γεωργία. Πιστεύω ότι το καθεστώς αυτό θα πρέπει να είναι παρόμοιο με αυτό των άλλων εργαζομένων. Συχνά, οι... αυτοί που λέμε ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι είναι ψεύτο αυτοαπασχολούμενοι, το ξέρουμε βρίσκονται σε καθεστώς ιονή μισθωτού. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουν παρόμοια δικαιώματα με αυτά των μισθωτών. Σε πολλές χώρες τα καθεστώτα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν προς το συμφέρον όλων να τροποποιηθεί η οδηγία αυτή και εν τέλει να τελειοποιηθεί θα έπρεπε η προσέγγιση αυτή να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζόμενους. Μισθωτούς, ανεξάρτητους, συζύγους ανεξαρτήτων. Παρέχει μια σειρά προτάσεων η συγγήτρια που προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του Συμβουλίου, κάτι θετικό. Ωστόσο, διαφωνώ λίγο μαζί της στο θέμα της μητρότητας. Πάλι για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και από την εισηγήτρια μεταξύ άλλων. Δεν δέχεται την θέση του Συμβουλίου να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών σε σχέση με τις μισθωτές ή ανεξάρτητες απασχολούμενες οι δύο ονόματι. Στη δεύτερη ανάγνωση πιστεύω ότι η θέση της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής πρέπει να είναι καλύτερη από αυτή που έχουμε υποβάλει στο δεύτερο τμήμα κύριο, Στο πρώτο, σωστά αναφέρθηκε, ότι η άδεια πρέπει να είναι ίδια, η διάρκεια δηλαδή της άδειας μητρότητας πρέπει να είναι ίδια με αυτή τη οδηγία του 92. Αλλά το δεύτερο τμήμα λέμε ότι ελπίζουμε να αλλάξει η οδηγία αυτή. Αφού δεν πήγε καλά μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει το Συμβούλιο βέβαια στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, καλό θα ήταν να υπογραμμίσουμε, και το θέλω, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να περιοριστεί στην παρουσίαση μιας έκθεσης, αλλά να παλέψει ούτως ώστε το Συμβούλιο να δεχθεί την εφαρμογή της νέας οδηγίας. Να μπορεί δηλαδή η οδηγία, ε, το καθεστώς να εφαρμόζεται και στις ανεξάρτητες, οι συζύγους ανεξαρτήτων ή ε, συντρόφους ανεξαρτήτων. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση του Συμβουλίου. Θεωρώ ωστόσο το ότι εφαρμο, ό,τι ισχύει για τη μία κατηγορία πρέπει να ισχύει και για την άλλη. Επαναλαμβάνω, συμφωνώ με το πρώτο τμήμα. Θα ήθελα ωστόσο στο δεύτερο τμήμα να πάμε λίγο πιο πέρα. Και με αυτή την οπτική θα ήθελα να αλλάξει και η τροπολογία 14 για να ευθυγραμμιστεί με την τροπολογία 5. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες νομίζω ότι μπορώ να τις δεχτώ εν πολλής, ε, βελτιώνουν εν πολλής τις θέσεις του Συμβουλίου. Εγώ θα ήθελα προφανώς να προχωρήσουμε παραπέρα στον υποχρεωτικό χαρακτήρα ενός μίνιμουμ κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των ε, εργαζομένων, είτε είναι αυτοαπασχολούμενες είτε όχι. Και βεβαίως και συζύγους. Στη γεωργία, στις υπηρεσίε στο εμπόδιο κλπ. Αυτό για να υπάρχει μία εγγύηση επαρκούς ενδεδειγμένου εισοδήματος για όλους τους πολίτες, για όλα τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με σεβασμό βεβαίως ε, της διαφορετικής κατάστασης που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, εξασφαλίζοντας ωστόσο ένα μίνιμουμ επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει νομίζω να αλλάξουν κάποια στοιχεία από αυτές ε, τις κυρίες Λού για να αναδεχθώ όλα τα άλλα. Η, κυρία, έχει, η κυρία Μωρά έχει δύο συγκεκριμένα αιτήματα που πολύ συχνά θέτει το έχουμε ακούσει πολλές φορές, μας έχει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Σας καλωσορίζω ε, και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό ανήκει στην παιδεία των παιδιών μας, των νέων πολιτών των Ευρωπαίων που θέλω να συμμετάσχω και γι' αυτό έχω πολλές ελπίδες ότι τελικά θα μπορέσουμε να ελέγξουμε σωστά το περιεχόμενο. Το έχω εμπιστοσύνη θα μπορέσουν να ελέγξουν οι παριστάμενοι την ε, εργασία τη Επιτροπής μας. Ευχαριστώ λοιπόν με τόσο καλοσύνη υποδεχτήκα τους φιλοξενούμενους μας. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής καταρχάς στο έργο της συναδέλφου μας Αστρίντ Λούλινγκ, η οποία αόκνος εργάστηκε επί του θέματος του δυσκόλου, ούτω ώστε και εδώ να επιτευχθεί πρόοδος και να βελτιωθεί η προστασία των γυναικών και οι συνθήκες εργασίας τους. Και ιδιαίτερα εδώ να προστατευθούν οι ανεξάρτητες εργαζόμενες. Συμφωνώ με αυτά που έλεγε η κυρία Χίλτα Φιγκερίδου. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι στις σημερινές μας εργασίες 25 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να προωθηθεί αυτή η κοινωνική προστασία των ε, ανεξαρτήτων γυναικών, των ανεξαρτήτων εργαζομένων. Οπότε εδώ έχουμε έναν καθήκον, πραγματικά καθήκον, να καταλήξουμε σε συμφωνίες, οι οποίες συμφωνίες θα είναι αποδεκτές της σπάση, διότι το ίδιο ισχύει και για τις συνθήκες που ισχύουν για τις εργαζόμενες. Κάτι για το οποίο προσπαθούμε. Συμφωνούμε τα υποθέτα. Υπάρχει πράγματι ανάγκη όλοι οι τομείς να καλύπτονται όσον αφορά τις ανεξάρτητες εργαζομένες. Η Κρίστα Κλάς μας είπε πόσο σημαντικό ήταν το θέμα για τις γεωργούς να καλύπτονται από αυτές τις διατάξεις. Αληθεύει όμως ότι όλες οι ανεξάρτητες εργαζόμενες και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, κυρίως στον τομέα της βιοτεχνίας, θα πρέπει και αυτοί να ωφεληθούν από αυτή την κάλυψη. Ευχαριστώ την Αστρίτ Λούλινγκ για το διαπραγματευτικό της πνεύμα, το γνωστό διαπραγματευτικό πνεύμα που επέδειξε, που επέτρεψε συνεργασία αγαστή με το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις διάφορες πολιτικές ομάδες και αναγνωρίζω το ότι άκουσε τη θέση διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων και της Γαλλίας, όσον αφορά ε, την τροπολογία 5 και πώς μεταλλάχθηκε αυτή. Η πρότασή της λοιπόν, επί της νέας διατυπώσεως της τροπολογίας 5, δεν μπορεί παρά να με χαροποιεί και την ευχαριστώ γι' αυτό. Παρομοίως, στην τροπολογία υπαριθμών θα ήθελα προφανώς να πω ότι καμιά φορά χρειάζονται ιδιαίτερες λύσεις, ειδικέ λύσεις που λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες, συγκεκριμένες περιορισμούς όσον αφορά την ανεξάρτητη εργασία. Είναι διαφορετική αυτή η εργασία από του μισθωτού. Και πιστεύω ότι εδώ μπορεί να υπάρξει συνάθρηση διαφορετικών εισοδημάτων. Όσον αφορά την άδεια μητρότητα, όσον αφορά τις ειδικές εισφορές μέσω των ειδικών εισφορών και διαφόρων εισφορών ε, και διαφόρων βοηθημάτων που μπορούν να δοθούν. Θα πρέπει να είναι πολύ ανοιχτή λοιπόν η τροπολογία που θα επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στα διάφορα κρατημέλη και οι ιδιαιτερότητες που είναι όλες εξίσου ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ την Astrid Λούλινγκ. Έχετε την εμπιστοσύνη μας κυρία Λούλινγκ για να ολοκληρώσετε τις διαπραγματεύσεις. Και έχετε την υποστήριξή μας στη δουλειά τη δύσκολη που κάνετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ο κύριος Όλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν κρατιέμαι. Θέλω να πω πως συμμερίζομαι τα σχόλια της κυρίας Φιγκερέδο όταν τονίζει πως ε, πραγματικά η κυρία Λούλινγκ σε αυτή την επιτροπή και η επιμονή που έχει επιδείξει στο να ενθαρρύνει την Κομισιόν ε, και τα άλλα θεσμικά όργανα μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα. Χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα και πρέπει να το πω αυτό. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφέρω ξεκάθαρα πως είναι ένα θαύμα το ότι έχουμε φτάσει σήμερα στη δεύτερη ανάγνωση. Μόλις πριν από ένα έτος ήμασταν στο Συμβούλιο να διαπραγματευτούμε αυτό το φάκελο και είχαμε πολύ μεγάλη αντίσταση. Όχι για τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για την ύπαρξη της οδηγίας εν μέσω της ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης. Γιατί συζητούσαμε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και έλεγαν τα κρατημέλη πως αυτό δεν είναι νόμιμο, είναι λάθος και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση από μεγάλα και μικρά κράτη-μέλη, ακόμα και για να το συζητήσουμε. Μέσω λοιπόν της δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Σουηδικής Προεδρίας καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο Συμβουλίο και όπως υπόθηκε η συμφωνία αυτή μπορούσε να είναι καλύτερη αλλά θα μπορούσε και να μην έχει υπάρξει καθόλου. Και ήταν πολύ λεπτή η διαφορά. Και η Κομισιόν υποστήριξε αυτή τη συμφωνία ε, γνώση του ότι εάν δεν την υποστήριζε δεν θα είχαμε κάποια συμφωνία γιατί χρειαζόταν ομοφωνία. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε αυτό κατά νου και με αυτά τα λόγια υποστηρίζω και την παρουσίαση της κυρίας Λούλιν πως είναι δύσκολος αυτός ο φάκελος και βεβαίως η Κομισιόν θα ήθελε να δει περισσότερα πράγματα από το Συμβούλιο πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα και να παραδεχτούμε πως δεν θα, θα πάρουμε πολύ περισσότερα ε, σκληρά λόγια αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας σήμερα οπότε συμφωνούμε με τις τροπολογίες της κυρίας Λούλινγκ σε μεγάλο βαθμό και με το σχέδιο έκθεση γιατί βελτιώνουν την έκθεση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν όλες στο Συμβούλιο, αλλά συμφωνούμε. Προσπαθούν να επιφέρουν σοβαρές βελτιώσεις και πράγματι υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να τονίσω κάποια πραγματάκια στη θέση του Συμβουλίου που είναι σημαντικά για να δείξουμε πως πραγματικά υπάρχει σοβαρή πρόοδος που γίνεται. Βεβαίω η παλαιά οδηγία του 86 δεν ε, μπορούσε να εφαρμοστεί. Ένας λόγος γι' αυτό που αφορούσε τις συζύγους που βοηθούν και την κοινωνική τους προστασία είναι το γεγονός ότι αν υπήρχε έμεση προστασία, έτσι ώστε να προστατεύονται μέσω του συζύγου ή σύζυγος, δεν υπήρχε υποχρέωση των κρατών μελών. Κάτι το οποίο πλέον έχει αλλάξει και είναι σημαντικό, γιατί μπορούμε άρα να εφαρμόσουμε την οδηγία, γιατί είναι σχεδόν πάντα έμεση προστασία. Αυτό το οποίο όμως θέλουμε και έχουμε τώρα, είναι άμεσο δικαίωμα για την σύζυγο η οποία βοηθά για την ίδια τη σύζυγο. Αμέσως και όχι Αυτό όνομα. Οπότε καλό είναι να μην κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση με την οδηγία 92 του 85 γιατί εδώ πέρα δεν πάμε από τις 14 εβδομάδες κάπου αλλού πάμε από το 0 στις 14 εβδομάδες που είναι και αυτό μεγάλη βελτίωση ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που είναι πιεσμένα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Να αναφέρω κάτι ακόμα που είμαι σίγουρος ότι θα εξηγήσει κατόπιν η κυρία Λούλινγκ καλύτερα από εμένα για αυτό το οποίο είπε η κυρία Τόμσον για την υποχρεωτική άδεια και για αυτό το οποίο είπε η κυρία Φιγκερέιδο για την οδηγία 92 του 85. Σημαντικό είναι εδώ πέρα, ειδικά όταν μιλάμε για άλλες κατηγορίες πλήν αγροτών, να εξετάσουμε τις πρακτικές συνέπειες του να μένουμε πάρα πολύ κοντά στην 92-85 στην άδεια μητρότητα. Εάν δούμε το ζήτημα πρακτικά, π.χ. μιας γυναίκας ιατρού. Εάν εφαρμόσουμε την 9285 θα έχουμε υποχρεωτική άδεια. Αυτό σημαίνει, θα έλεγα εγώ ως δικηγόρος, πως αυτή η γιατρός δεν μπορεί να δει καν τα email της κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και είναι σε διαφορετική θέση από έναν υπάλληλο, γιατί μπορεί να χάσει πολλούς πελάτες, γιατί δεν μπορεί να ασχοληθεί με κανένα θέμα της ε, δουλειάς της π.χ. κατά τη διάρκεια της άδεια. Οπότε πρέπει να δούμε το τι σημαίνει αυτό πραγματικά, δηλαδή το να κινηθούμε πάρα πολύ κοντά στην 92 του 85, γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση. Και Ε, θα οδηγηθούμε σε κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά το νόμο που θα εφαρμόζεται. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως υπάρχει ο φορέας ε, της ισότητας ε, και η δυνατότητα συνδέσμων ενώσεων που θα μπορούν να πηγαίνουν στα δικαστήρια εξ των μελών τους, ξεκάθαροι κανόνες για αποζημιώσεις και ένα άρθρο ρητά που επιτρέπει την θετική δράση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα των γυναικών, την οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υποστηρίξουμε την γυναική επιχειρηματικότητα γιατί είναι πολύ χαμηλά τα νούμερα. Δεν θέλω λοιπόν να σφάλω χρόνο. Στηρίζω πλήρως το σχέδιο έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Όλσον. Για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα και πολύ εποφελή συζήτηση, δίνω ξανά το λόγο στην εισηγήτρια. Κυρία Λούλινγκ. Ε, ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους όσοι μίλησαν, όσες μίλησαν μάλλον στη συζήτηση. Με την κυρία Κλά σύμφωνα απόλυτα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Κύριε Τόμψεν, είναι σαφές ότι το πεδίο εφαρμογή δεν περιορίζεται πλέον διότι το Συμβούλιο δέχθηκε πλήρως την τροπολογία μας είχε κρατήσει την οδηγία, αλλά δεν είχε ενημερωθεί σωστά. Στην άλλη τροπολογία όμως λέγαμε ότι η νέα αυτή προστασία πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση των ανεξαρτήτων εργαζομένων και των, των γυναικών ανεξαρτήτων εργαζομένων και των συζύγων ανεξαρτήτων εργαζομένων. Δεν αναφέρουμε πλέον κανένα τομέα, άρα προφανώς καλύπτονται όλοι οι κλάδοι το εμπόριο, η βιοτεχνία, τα ελεύθερα επαγγέλματα. Στη χώρα μου υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί γιατροί, οι γυναίκες των οποίων κάνουν το γραμματέα των γιατρών. Οι γιατροί είναι ανεξάρτητοι στη χώρα μου. Άρα καλύπτονται οι πάντες. Κανένα ανεξάρτητο εργαζόμενο σε κανένα τομέα δεν υπάρχει που να μην καλύπτεται με το κείμενο τη τροπολογία μα, επί του οποίου συμφώνησε το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικαίωμα να αφαιρείς από τη φορολογική σου δήλωση τις εισφορές, γιατί κανονικά πληρώνεις εισφορές. Στους μισθωτούς πληρώνει ο μισθωτός και ο εργοδότης. Εμείς προτείνουμε μια μεγάλη τροπολογία για το δικαίωμα αφαίρεσης ε, του φόρου της εισφοράς. Τη ε, επαγγελματική φορά. Εδώ δεν συμφωνεί το Συμβούλιο, αλλά πρέπει να σα πω ότι το πρόβλημα αυτό ε, ε, βαθιά την αρχή της επικουρικότητας. Το κράτο πρέπει να είναι αυτό που θα αποφασίσει αν μπορεί ε, να δεχτεί ή όχι να αφαιρούν, να εκπίπτουν του φόρου τις, ε, οι σφορές. δική μου χώρα αυτό έχει ισχύσει, στη Γεωργία και αλλού όλοι ε, οι ανεξάρτητοι σε εμά και οι σύζυγοι ανεξάρτητων τίσουν παρέκκληση είναι ε, εγγεγραμμένοι. Αλλά προφανώς αφαιρούνται οι εισφορές τους από το φόρο όπως οι εισφορές των μισθωτών. Αλλά αυτό είναι θέμα που θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό δεν το χρειαζόμαστε στην πράξη να το αναφέρουμε εδώ. Τώρα, για την υποχρεωτική διάρκεια της μητρότητας θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε υποχρεωτική άδεια σε ανεξάρτητους. Δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό. Αυτοί θα αποφασίσουν. Πόσο καιρό θέλουν και είναι πολύ δύσκολο να πεις σε ένα γιατρό ότι, σε μία γιατρό ότι δεν μπορείς να δέχεσαι ασθενείς για μία χύπη χρονική περίοδο. Και νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζεται να αναφέρουμε για την υποχρέωση αυτή, άλλωστε το κοινοβούλιο δεν το έχει ζητήσει. Σε ό,τι αφορά τον φορέα, ξεκάθαρη είναι η θέση μας, ο ίδιος φορέας με αυτόν που αντιμετωπίζει την αρχή ισότητας ε, των μισθών στον τομέα των μισθωτών. Για την κυρία Φιγκερέδο, την ευχαριστώ όντως 20 χρόνια συνεχώς το ζητάγα, το ζήταγε να, ζητάγαμε να αλλάξει η οδηγία του 86 δεδομένης της ηλικία μου να πω της Κομισιόν ότι δεν θα σας ε, κυνηγάω άλλα 20 χρόνια, αλλά χαίρομαι που μπορώ να θέσω πέρα σε αυτή την παρενόχληση. 5-10 χρόνια τώρα δεν ξέρω, μπορεί. Για το πεδίο εφαρμογής είναι σαφές, το είπα, αφορά όλες τις ε, ανεξάρτητες, συμφωνεί το Συμβούλιο. Όλα βεβαίως εξαρτώνται από το καθεστώς που έχουν οι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι στα κράτη-μέλη. Εμεί ζητάμε την ίδια προστασία για το σύζυγο, όπως και για τον ίδιο τον ανεξάρτητο εργαζόμενο. Πλην όμως, το καθεστώς από χώρα σε χώρα διαφέρει. Η οδηγία πάει μακριά τουλάχιστον έτσι όπως είναι το πνεύμα του Συμβουλίου. Δεν μπορώ να τους αλλάξω. Είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι ήταν μικρό θαύμα αυτό. Ξέρω τι έγινε στις συζητήσεις του Συμβουλίου. Εγώ θα ήθελα να είναι λίγο μεγαλύτερο το θαύμα, αλλά η κατάσταση είναι πολύ ευέλικτη. Κάποια μέλη του Συμβουλίου λέ, θέλανε να πούν υπάρχει κρίση για να μην ε, περάσουν, να μην γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι καλό είναι να κλείσουμε την κατάσταση τώρα και να περάσει η οδηγία στη δεύτερη ανάγνωση με τις τροπολογίες που προτείνουμε και είμαι βέβαιο θα το πετύχουμε. Για τη μητρότητα, είπε η κυρία Φιγκερέντο ότι σα ασφαλισμένου αυτό έχει διαφορετική άποψη. Να σας πω εγώ το εξή όμω. Εμεί στην οδηγία αυτή δεν μπορούμε να ζητήσουμε να υπάρχουν πράγματα που δεν δέχεται η άλλη οδηγία. Και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει κάτι τέτοιο. έχουμε προχωρήσει από τις 0 στις 14 εβδομάδες. Υπάρχει ένα κείμενο που λέει σαφώς ότι όταν η διάρκεια μητρότητας των μισθωτών αλλάξει, η Κομισιόν θα υποβάλει έκθεση για προσαρμογή της οδηγίας. Ε, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα από, από εδώ, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε εδώ και τώρα πράγματα που δεν είναι σαφή είναι που είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι το κείμενο που προτείνω πάει αρκετά μακριά. Ελπίζω να πείσω το Συμβούλιο και εγώ θα προτιμούσα να πάω πιο μακριά. Κύριε Μωρά, ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να φέρω κοριτσάκι εδώ, δεν έχω. Θα μπορούσα να σας φέρω ε, μικρανεψιές μου αν θέλετε, για να σας κάνω ανταγωνισμό. Εγγονές δεν έχω. Για την τοπολογία 15 και 11. Είχα επαφή με την ε, μεγαλική με τη γαλλική αντιπροσωπεία. Θα βρούμε ένα σωστό κείμενο για την γλωσσική εκδοχή. Θα ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, διότι η περικοσαετής παρενόχλησή μου απέδωσε. Κράτησε, δεν ήταν εύκολη, αλλά ξέρετε, εγώ δεν τα παρατάω. Συνεχίζω και ξέρετε δεν ήταν σεξουαλική παρενόχληση, ήταν και διανοητική. Είπα ότι θα υποσχεθώ στην Επιτροπή να μην συνεχίσω την παρενόχληση την επόμενη 20 ετία, αλλά σίγουρα θα έχω κάποιον διάδοχο. Και ευχαριστώ την Επιτροπή που εν τέλει υπέβαλε μια πρόταση οδηγία και ευχαριστώ που συνέβαλε στην διαμόρφωση αυτού του μικρού θαύματος στο Συμβούλιο που επέτυχε αυτή την κοινή θέση κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θα δω τις τροπολογίες και θα διαπραγματευτούμε για να υπέλθει μια συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Και ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ. Όλοι μας. Ελπίζουμε πράγματι αυτή η προσπάθεια να στεφτεί με επιτυχία. Διότι πραγματικά κατελήσαμε μεγάλες προσπάθειες. Και τα αποτελέσματα τα σωστά θα είναι πολύ θετικά για τους ανεξάρτητες εργαζόμενες και για τους συζύγους. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 8 Απριλίου στις 5 το απόγευμα. Αύριο ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Γυναικών, 3 και 4 Μαΐου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια στη δεύτερη, το Μάιο, στη σύνοδο του Στρασβούργου το Μάιο. Κλείνουμε εδώ αυτό το σημείο και πάμε στο επόμενο. Έκθεση Φιγκερέιδο όσον αφορά τα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον. Όσον αφορά αυτό το θέμα, θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Φιγκουερέιδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το... Αυτή είναι μια δεύτερη συζήτηση που διεξάγεται. Επί μιας εκθέσεως που αφορά τα αποτέλεσμα αυτού του οδικού χάρτη για την ισότητα ανδρών και γυναικών 2006-2010 και τις συστάσεις για το μέλλον. Και μετά από κάποιες αντιρρήσεις που προευλήθησαν από πλευράς ΕΛΚ κυρίως και μετά από μια συμφωνία που επετεύχθη τελικά διαφαίνεται μια δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Θέλουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Αυτή η έκθεση πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας. Δηλαδή να έχουμε μια μελλοντική στρατηγική για την ισοτιμία ανδρών γυναικών. Πιστεύω λοιπόν ότι βασιζόμαστε και στην πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοίνωσε η κυρία Ρέντινγκ ότι το Σεπτέμβριο θα υποβληθεί νέα πρόταση. Και ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα θεωρηθεί ως μια συνεισφορά στην πρόταση της κυρίας Ρέντινγκ. Όπως είπα, εμείς μέσω της εκθέσεως θέλαμε να πετύχουμε ευρία συνένεση στο Κοινοβούλιο και να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία που θα υποστηρίζει ε, την έκθεση αυτή στην επόμενη Ολομέλεια. Στο σχέδιο εκθέσεως έλαβα υπόψη διάφορα θέματα που εθίγησαν από τα μέλη, διάφορα ζητήματα, αρκετά μέλη έκαναν δικές τους προτάσεις που συμπλήρωναν το σχέδιο εκθέσεως também Όπως γνωρίζετε, το μήκος της εκθέσεως περιορίζεται και σε πρώτερη συζήτηση είπα ότι δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω όλες τις ιδέες που ήθελα. Όμως έχουμε 7 νέες προτάσεις και έκανα κάποιες αλλαγές στο σχέδιο της έκθεσης. και νομίζω ότι οι προτάσεις και οι αλλαγές, αν συμπεριληφθούν στην έκθεση, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πετύχουμε τη συνένεση. Έχουμε νέα, λοιπόν τροπολογίες, οι 8 και 9 είναι οι δικές μου τροπολογίες που αφορούν την παράγραφο 11 και την παράγραφο 17 του σχεδίου κειμένου, του σχεδίου της εκθέσεως. Οι άλλες προτάσεις που υπευλήθησαν για νέα στοιχεία προς συμπερίληψη ή στην έκθεση. Οι προτάσεις αυτές, λέω, αφορούν τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Αν δείτε αυτές τις τροπολογίες που προανέφερα, θα δείτε ότι εν λόγω τροπολογίες περιγράφουν διάφορες θέσεις θέσεις οι οποίες αναφέρονται στον οδικό χάρτη 2006-2010 στον οδικό χάρτη αυτό που συζητούμε. Και ο οδικός χάρτης αυτός καλύπτει έξι βασικά θέματα, οικονομικά θέματα, απασχόληση, αμοιβέ μισθούς. Αυτές οι τροπολογίες αναφέρουν ότι έχουν επιτευχθεί κάποιες πρόοδοι, αλλά μόνο περιορισμένες. Είναι περιορισμένη η πρόοδος. Και γι' αυτό αναφέρεται ότι θα πρέπει τώρα να γίνουν νέες προτάσεις, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι ανισότητες που υπάρχουν στην απασχόληση, να μειωθούν οι διακρίσεις όσον αφορά τις αμοιβέ στην τροπολογία 3. Εκεί αναφερόμαστε στην συμφιλίωση της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής με την επαγγελματική ζωή. Επίσης, η τροπολογία συγκεκριμένη αναφέρεται στην μητρική πατρική άδεια και ούτω καθεξής, στη γονική άδεια. Και η τροπολογία αναφέρει ότι εδώ απομένουν πολλά να γίνουν. Η τροπολογία 4. Εδώ στην τροπολογία 4 έχουμε αναφορά στη συνεχιζόμενη διάκριση όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στην οικονομική ζωή και στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και στην πολιτική ζωή. Στο σημείο 5 αναφερόμαστε στο Δάφνη 3, πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, προφανώς, και λέμε ότι περαιτέρω μέτρα απαιτούνται ούτω ώστε να εκριζωθεί η βία μεταξύ των φίλων. Μετά έχουμε τροπολογία 6. Εκεί αναφερόμαστε στη συμπερίληψη της ισότητας των φίλων ως προτεραιότητας στην παιδεία, στην κοινότητα, στα προγράμματα κατάρτισης και παιδείας, ούτως ώστε να μειωθούν τα στερεότυπα στην κοινωνία και πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα. Αυτό αναφέρεται εδώ. Και λέμε ότι χρειάζονται και άλλες προτάσεις. Στην τροπολογία 7, εδώ αναφερόμαστε στη στις δηλώσεις, διακήρυξη των στόχων της χιλιετίας και της ειδικής πλατφόρμας επί της οποίας βασίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει δεσμευθεί να ακολουθήσει αυτές τις αρχές. Και στο τέλος της εκθέσεως αυτές οι αρχές αναφέρονται εκτενέστερα. Όπως προανέφερα, οι τροπολογίες 8 και η τροπολογία 9 είναι τροπολογίες δικές μου, αφορούν το αρχικό κείμενο. Στην τροπολογία 8 αποσύρω την αναφορά μου στους 12 τομείς που καλύπτονται διότι στις πρώτερες έξι τροπολογίες αυτοί το τομείς καλύπτονται. Γυναίκες και φτώχεια, παιδεία και κατάρτιση των γυναικών, γυναίκες και υγεία κλπ. κλπ. Επίσης, δέχομαι ότι αυτά τα σημεία καλύπτονται στον οδικό χάρτη, στο χάρτη πορείας. Έχουμε τροπολογία 9 μετά. που αναφέρεται στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Εδώ ήθελα να αναφέρομαι γενικόλαγα σε αυτά και ραπέμπω σε πρώτερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα πάντα εδώ, στην παράγραφο 17, αναφέρονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αυτό είναι το πιο πρόσφατο κείμενο της έκθεσης. Σκιαγράφησα πιστεύω τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί που θα μας δώσουν τη δυνατότητα πιστεύω να ετοιμαστούμε για το υπόλοιπο της συζητήσεως. Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε και άλλες τροπολογίες, έχετε χρόνο μέχρι τις 9 του μηνός. Άρα είναι ευπρόσδεκτες τυχόν τροπολογίες μέχρι τότε. Έχουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την έκθεση, κάτι που συμφωνήσαμε στη συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα η συζήτηση του σχεδίου Έκθεση Πρώτα απ' κυρία Γκόμες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε. Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν που προσκάλεσε διάφορους συμμετέχοντες στις διάφορες επιτροπές και ειδικά όσους είχαν συνεισφέρουν από την Επιτροπή Άμυνα. θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίγκερέιδο για το εξαιρετό έργο της και καλωσορίζω κάποιες από τις αλλαγές που έκανε στο σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να την ευχαριστήσω που δέχτηκε και κάποιες τροπολογίες τις οποίες ε, εξήγησε κιόλας. Νομίζω πως η έκθεση είναι επίκαιρη. Είναι μια απαραίτητη συνεισφορά στην ε, πρόταση της Κομισιόν που προετοιμάζει η κυρία Ρέντινγκ και θα συνεισφέρει γενικά στην ισότητα, στρατηγική ισότητα μεταξύ των φύλων και στα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά, όσον αφορά τις γυναίκες. Επίσης, ε, συμφωνώ πλήρως ε, με τις προτάσεις της κυρίας ε, Φιγκερέιδο για μια ετήσια τριμερή συνάντηση και για μια διάσκεψη που θα πρέπει να γίνεται για την ισότητα των δύο φύλων και θα πρέπει να οργανώνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το βασικό μας θέμα εδώ πέρα είναι οι δείκτες. Νομίζω πως είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε κάποιους δείκτες που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να παρακολουθούμε την κατάσταση των γυναικών. Τώρα, για να ξαναδούμε την δική μου εμπειρία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Εγώ θα προετοιμάσω κάποιες ε, τροπολογίες εντός της ε, προθεσμίας και επί τη ευκαιρία στο σημείο 7 γίνεται λόγος ε, για το έργο των σχετικών γενικών διευθύνσεων στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο και για τη δουλειά που θα πρέπει να κάνουν στον ε, τομέα της ισότητας των δύο φίλων. Νομίζω πως αυτό θα είναι σημαντικό κομμάτι της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουν το θέμα της ισότητας. Και νομίζω πως θα είναι καλή ιδέα να το υπογραμμίσουμε αυτό σε αυτήν εδώ την έκθεση. Βεβαίω, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση των γυναικών στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Θυμάμαι πως ε, όταν είχα γράψει εγώ τη σχετική έκθεση το 2007 καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως υπήρχε δυσαναλογία στον αριθμό των γυναικών που απασχολούνταν σε θέσεις λήψης αποφάσεων και δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα έκτοτε. Οπότε νομίζω πως πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μια προσπάθεια για να υπάρξει περισσότερη ισότητα στα ίδια τα θεσμικά όργανα. Οι τροπολογίες 8 και 9 τώρα τις παραγράφους 11 και 12 της έκθεσης. Αναφέρουμε εδώ ρητά ότι πρέπει να υπάρχουν πρακτικές εφαρμογές της ισότητας που να αφορούν κάθε διάσταση της πολιτικής και εξωτερική πολιτική. Να τονίσω επίσης και μια άλλη μνήμα που έγινε στους στόχους της χιλιετίας του ΟΗΕ. Πρέπει να αναφερόμαστε σε πολιτικές που θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ισχύ στις γυναίκες. Βεβαίως να αναλάβουμε πρωτοβουλίες στο Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση τέτοιων πρωτοβουλίων, αλλά πρέπει η έκθεση να το αναφέρει και ρητά. Επίσης, ε, πρέπει να κάνουμε Μενία και στη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας με τη νέα συνθήκη. Η πολιτική ωστόσο θα πρέπει, η πολιτική μας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται παρκώς υπόψη οι θέσεις των γυναικών όταν διαμορφώνονται εξωτερικές πολιτικές ή αμυντικές πολιτικές της Ένωσης. Κάτι επίσης θα έπρεπε να τονίσω είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν το ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ένα ψήφισμα για το ρόλο των ειρηνικών δραστηριοτήτων, των ειρηνικών αποστολών. Πιστεύω και στον τομέα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούμε την, ε, να συμπεριλάβουμε το ρόλο των γυναικών εκεί. Ως προς τα λοιπά, απλά να συγχαρώ την εισηγήτρια. Δυστυχώς η, η άλλη εισηγήτρια δεν μπορεί να είναι παρούσα, διότι βλέπετε πολύ σημαντικέ γυναίκε στην ομάδα μου, τη ζητούν παντού και είναι συνάδελφο στην Νορβηγία, η Γκόντερ, και τη υποσχέθηκα να διαβάσω την συνεισφορά τη στη συζήτηση. Ξεκινώ την ανάγνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Λόγω των ανηλυμένων μου υποχρεώσεων λυπούμε που δεν μπορώ να παρίσταμαι στη συζήτηση τη πολύ σημαντική αυτή εκθέσεω. Καταρχά, πρέπει να πω ότι είμαι ικανοποιημένη που είμαστε πιο κοντά σε συμβιβασμό τώρα από ότι ήμασταν πριν από τρει εβδομάδε. Η Ιλντα Κολ το θεωρεί ότι αυτό είναι συνένεση. Ευχαριστώ τους, ε, την κυρία Φιγκουερέιδο που ήταν τόσο συνεργάσιμη και τόσο ανοιχτή συζητήσει. Νομίζω ότι οι νέε εννέα τροπολογίε αντιπροσωπεύουν σοβαρή προσπάθεια αξιολόγηση των επιτευχθέντων μέσω του οδικού χάρτη 2006-2010 για την ισότητα των φύλων. Όμω ε, υπάρχουν κάποια σημεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Να περιγράψω ακροθυγώ τι πρώτερε τροπολογίε μου. Πρώτα απ' όλα θέλω να είμαστε πιο ευθύ όσον αφορά του πόρου. Αν θέλουμε συγκεκριμένε δράσει, συγκεκριμένε πολιτικέ, και αν καταλαβαίνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό επιθυμούμε, εδώ χρειαζόμαστε πόρους. Ε, επί μακρόν, έλεγα ότι ο δικός χάρτης θα πρέπει να εμπεριέχει στόχους και να τη στόχη από τους πόρους. Πιστεύω ότι αυτό χρειαζόμαστε. Επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους ισότητας των φύλων ε, που θα συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές ε, που θα προτείνει θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναλύσουν τα διάφορα προγράμματα για την καταπολέμηση της κρίσεως και εξόδου από την κρίση από την γυναική άποψη. Υπέβαλα μια τροπολογία σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις γνωρίζοντας ότι πρόκειται περί θέματος που επιδεινώνει τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών στην Ευρώπη. Τις επόμενες μέρες θα υποβάλω μία-δύο ακόμα τροπολογίες που θα ήθελα η Επιτροπή να συζητήσει. Η πρώτη αφορά το πρόβλημα της διαφοράς μεταξύ των αμοιβών και ενδεχόμενες πολιτικές καταπολέμησης αυτών. Δεύτερον θέμα θα είναι η πρόκληση ε, της χάρτας δικαιωμάτων της γυναίκας. Ο πρόεδρος Μπαρόσο και η επίτροπο Ρέντινγκ ήδη εξέδωσαν ένα σχέδιο κειμένου και νομίζω ότι η Επιτροπή Γυναικών θα πρέπει να επιμείνει στη συμμετοχή της για περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τέλο παράθεση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τόμσον. Ευχαριστώ κυρία Λαρούσοβα τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Φιγκέρεντο για την έκθεσή της. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια βούληση να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις, τις υποστηρίζω. Ωστόσο νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορούν ακόμα να ε, προωθήσουν. Θα, θα είμαι σύντομη. Θέλω απλά να υπογραμμίσω τρία σημεία. Πρώτον, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ισότητα Ανδρών Γυναικών. Αυτό θα, το Ινστιτούτο θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη ε, παρουσία αν επικαιροποιούσε τους δείκτες. Φροντίστε λοιπόν οι δείκτες αυτοί να με τους στόχους που θέσαμε εξ αρχής. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε ευκολότερα να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Κατόπιν, όταν μιλούμε για εσωτερική λειτουργία, πρώτον, της Γενικής Διεύθυνσης επιτροπή, μην ξεχνάτε ωστόσο ότι μέσα στους ε, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι σημαντικό να υπάρχουν ή να εισαχθούν ε, ενισχυμένοι μηχανισμοί συντονισμού, να υπάρχει συνέχεια και να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα με βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμους στόχους που θα αναθεωρούνται κάθε χρόνο. Επίσης, θα πρέπει από τη μια μεριά να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα, αλλά από την άλλη να προωθήσουμε τις βέλτισες πρακτικές. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν εκστρατείες ε, ευαισθητοποίησης. Εν ολίγης, θα έλεγα ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η, τοπική, η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές δομές πρέπει να έχουν μια συνεκτική ενοποιημένη προσέγγιση. Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε η συγγήτρια μα επέτρεψε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης συνολικά. Ευχαριστώ κύριε Νεντάρσεβα. Η κυρία Γκαρσία Πέρε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Επαναλαμβάνω και εγώ τις ευχαριστίες μου για την ε, κυρία Φιγκερέδο για την έκθεσή της να κάνω μια πιο γενική παρατήρηση. Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, ε, κάποιες περιπτώσεις μάλλον, όπου ε, λέγεται ότι στην Επιτροπή Γυναικών, στις γενικές ε, συζητήσεις, επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα σε ό,τι αφορά την ισότητα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος, να μην συνεχίσουμε να θέτουμε τα ζητήματα αυτά και να επιμένουμε στα ζητήματα αυτά. Και το λέω γιατί, διότι πιστεύω ότι οι τελευταίες, στις τελευταίες παρατηρήσεις υπήρχαν ορισμένες κάτι που μερικές φορές ξεχάστηκε ή δεν ξέρω αν είναι εσκεμμένο ή όχι, στο να αναφέρονται οι διαστάσεις φύλου σε κάποιες ε, ευρωπαϊκές πολιτικές. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να πρέπει να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε σαφείς στόχους όπως την ανάγκη να ενσωματώσουμε τη γυναίκα στην αγορά εργασία, να, να, γίνει, να, να, να, υπάρξει, να αντιμετωπιστεί οι, οι μισθολογικές διαφορές. Αυτά είναι θέματα που, επαναλύ, που συζητήθηκαν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να τα λέμε, να Άλλο σημαντικό ζήτημα. Η έμφυλη βία. Η μάχη κατά της έμφυλη βία είναι πολύ σημαντική στις κοινοτικέ πολιτικές, σε όλο το θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επιμένουμε στους στόχους αυτούς. Η στρατηγική Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020 πρέπει σαφώς να έχει και μια έμφυλη διάσταση, με συγκεκριμένες θέσεις, συμμετοχή της γυναίκας στην ε, αγορά εργασία, μάχη κατά των μισθολογικών ανισοτήτων, με συγκεκριμένους στόχους που θα επιβάλλουν στα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα να θέσουν σε κίνηση όλα τα αναγκαία εργαλεία για να προχωρήσουμε στην αρχή της ισότητας. Με ευχαριστώ, κύριε Γκρασία Πέρες. Η κυρία Μπάουερ έχει τώρα το λόγο. Mm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα αναφέρω κάτι ελαφρώς διαφορετικό από αυτά τα οποία συζητάμε. Αναγνωρίζω πως η κυρία Φιγκερέδο είναι πολύ εργατική ευρωβουλευτής και εργάζεται ταυτόχρονα σε πολλές εκθέσεις και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ορισμένες φορές όμως έχω την αίσθηση πως ε, χάνουμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω πως αυτό συμβαίνει τώρα όταν πρέπει να και όταν θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, αντί να σταματήσουμε λίγο και να δούμε τι δουλεύει και τι δεν λειτουργεί. Και νομίζω πως η ε, έκθεση αυτή είναι μια ευκαιρία να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το οδικό χάρτη 2006-2010. Πώς δουλεύει, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους δεν ε, λειτουργήσε κτλ. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως υπάρχει μια έλλειψη υπομονής. Εντάξει, αυτό ισχύει για όλους μας, όλοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα αντί να μιλάμε για το παρελθόν δεν είναι τόσο συναρπαστικό να κοιτάμε συνεχώς το παρελθόν, αλλά εάν δεν δούμε το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, τι είναι αποτελεσματικό και τι δεν είναι αποτελεσματικό, εάν δεν δούμε πού έχουν μειωθεί και πού έχουν αυξηθεί οι ανισότητες, τότε δεν θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε τους σωστούς στόχους. Οπότε νομίζω ότι τρέχουμε πολύ γρήγορα κάποιες φορές, γιαζόμαστε πάρα πολύ και οι τροπολογίες φαίνεται πως αποκαθιστούν κάπως αυτή την ισορροπία. Θεωρώ παρόλα αυτά πως δεν θα πρέπει να γράψουμε μια έκθεση για το τι θα θέλαμε να επιτύχουμε στο μέλλον. Δεν πρέπει να αφορά μόνο στόχους, Αντιθέτως η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει και το ποια ήταν εκείνα τα πράγματα τα οποία λειτουργήσαν και αυτά τα οποία δεν λειτουργήσαν σε αυτή την ε, περίοδο, στην περίοδο του οδικού χάρτη, ποιοι ήταν οι αποτελεσματικοί παράγοντες, ε, ποια ήταν τα πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Πιστεύω πως θα ήταν καλή ιδέα να αναφέρουμε τις έξι προτεραιότητες, να αξιολογήσουμε το τι έχει γίνει, το τι δεν έχει γίνει, τι ήταν αποτελεσματικό και τι όχι. Είμαι σίγουρος πως το Ινστιτούτο των φίλων είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά και θέλω να είμαι προσεκτική εδώ πέρα, δεδομένου του ότι δεν είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της ε, έκθεσης, Φαίνεται πως εδώ πέρα εστιάζουμε στο τι θα έπρεπε να συμβαίνει. Και δυσκολεύομαι λίγο εδώ πέρα. Φαίνεται πως κάποια από τα... Ε, δεν υπάρχει η βάση απαραίτητη για το, στην έκθεση για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Δεν νομίζω λοιπόν πως και οι έξι αυτές τροπολογίες ε, μπόρεσαν να αποκαταστήσουν την ισορροπία που χρειαζόμαστε. Και βεβαίω δεν θέλω να εκλειφθεί αυτό ε, προσωπικό σχόλιο. Όλοι φταίμε γι' αυτό. Μας αρέσει να κοιτάμε το μέλλον. Έχουμε εμπειρίες, έχω προσωπικές εμπειρίες για το χάσμα το μισθολογικό. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, ε, που είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ποιες είναι οι δράσεις ε, που μπορούμε να αναλάβουμε. Θεωρώ λοιπόν πως η όλη αυτή η έκθεση δεν ε, κάνει αυτή την αναδρομή για να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να ξαναδείτε την έκθεση από αυτό το φως για να μην χάσουμε και αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Οβίρ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να συνεχίσω εγώ από εκεί που σταμάτησε η κυρία Μπάουερ, αλλά πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Φιγκερέδο, γιατί πραγματικά έγραψε μια έκθεση κοιτώντα στο μέλλον. Και με ειλικρίνη, αλλά νομίζω πως χρειαζόμαστε εδώ πέρα μια νέα όθηση. Έχουμε ακούσει πολλές καλές σκέψεις όλα αυτά τα χρόνια, είτε φορούν τη βία, είτε φορούν την πληρωμή. Είναι ζητήματα μας απασχολούν δύο-τρεις ε, δεκαετίες, αλλά σε έναν κόσμο με κέντρο τους άντρες δεν υπάρχει θέληση να λάβουμε μέτρα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως το χάσμα των μισθών αυξάνεται. Το 2007 ήταν 17% αντί για 14% και η ανάλυση για το 2009 μας δείχνει πως η ψαλίδα και πάλι θα ανοίξει. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την προσέγγισή μας και να αγωνιστούμε για τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεων μας. Έχουμε γράψει συντάξει πολλά καλά έγγραφα, αλλά η Κομισιόν που έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι δεν έχει αναλύσει γιατί κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν λάβει μέτρα για να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών ή την ψαλίδα στις αμοιβέ ή το γιατί η εκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα είναι τόσο χαμηλή. Είναι σαφές πως ε, δεν έχουν λειτουργήσει λοιπόν αυτά τα μέτρα. Χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση και δεύτερον όλες αυτές οι σκέψεις είναι σωστές που αναφέρονται στα έγγραφά μας. Τι λείπει όμως, λείπει ένας μηχανισμός επιβολής και επιτήρησης. Χωρίς αυτά τα μέτρα μας δεν θα λειτουργήσουν όπως θέλουμε τις ε, επόμενες δεκαετίες. Συνελώνται οι πίν λοιπόν. Βλάπτει αυτό την συνείδηση της κοινωνίας το να μην εφαρμόζονται οι νόμοι. Ευχαριστώ κύριε Οβίρ. Η κυρία Μπρινκεβισιούτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κυρία Φιγκερέντο, για την έκθεσή της. Γιατί για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον πρέπει να μπορούμε να αναλύσουμε το παρελθόν. Ωστόσο, δεν θα έχουμε και το χρόνο για την ανάλυση αυτή. Νομίζω ότι αποφύ, αποτύχαμε να εφαρμόσουμε τις προηγούμενες οδηγίες και τις προηγούμενες καθηγητές γραμμές, συγγνώμη, για την ισότητα και μπορεί να χρειαστεί να ψάξουμε να βρούμε τι πήγε λάθος, ποιος έφταιγε. Μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική κατάσταση έπαιξε ρόλο, η φτώχεια αυξήθηκε σε κράτη-μέλη, δεν μειώθηκε. Τώρα τι γίνεται. Η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού είναι επαρκής για να καταπολεμηθεί η φτώχεια πραγματικά. Μήπως είναι καιρός να περάσουμε σε μια οδηγία για ελάχιστα κοινωνικά στάνταρτ. Κατά την άποψή μου, μόνο μια τέτοια οδηγία θα μας δώσει τη δύναμη να χτυπήσουμε τη φτώχεια σε πραγματικά μεγέθη στα κράτη-μέλη. Και παρεμπιπτόντος, η φτώχεια πλήττει τις γυναίκες περισσότερο, ιδίως τώρα μετά την ύφεση. Τώρα στη φάση της ύφεσης οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα περισσότερα μειονεκτήματα. Η μισθολογικής ανισότητας λόγω ε, φύλου επιδεινώνονται και νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αλλάξει την οδηγία για τους μισθούς. Αν δεν έχουμε μια καλή οδηγία για τα επίπεδα μισθών, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση με αναφορά καλών παραδειγμάτων σε κάποια κράτη-μέλη. Ένα άλλο πρόβλημα. Αυξάνεται η βία κατά των γυναικών και η διακίνηση γυναικών. Και εδώ θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να υιοθετήσουμε μέτρα που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Να συγχαρώ εκ νέου την εισηγήτρια. Μετά τις συζητήσεις πρέπει να λάβουμε απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μπρινκεβιτσιούτε. Έχει και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να πει κάτι. Η κυρία Φίνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Στρέλλα που μας δίνεται εντάχει την ευκαιρία να συγχαρώ την κυρία Φιγκερέντο για το σχέδιο έκθεσης που αποτελέζει μια πολύ διαφορετική βάση για την Επιτροπή εν ώψη της προετοιμασίας της νέας στρατηγικής μας. Να σας υπενθυμίσω εντάχει ότι η νέα στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών θα παρουσιαστεί μετά την έκκριση της χάρτας που εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου. Η στρατηγική αυτή θα επικεντρώνεται σε δεσμεύσεις που θα λάβει η Επιτροπή για την εντολή της και θα αφορά δράσεις που θέλει να υιοθετήσει για την περίοδο του 2010 στο 2015. Να σας επιβεβαιώσω λοιπόν ότι προβλέπεται να εγκριθεί η στρατηγική το Σεπτέμβριο και ότι χρειάζεται στην αυτή στρατηγική να υποβάλουμε τις, να παρουσιάσουμε τις αρχές που αναφέρθηκαν στο χάρτη των γυναικών και που αντιστοιχούν εν γέννη στους βασικούς τομείς που υπογράμμισε η έκθεση που παρουσιάζεται και σήμερα. Επιπλέον, πέραν των τομέων που θα καλύπτει η στρατηγική εν γέννη, θα υπάρχει και μια έμφαση που θα αφορά όλες τις διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της διακυβέρνησης του τομέα ισότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιμο να επενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή θέλει να ενισχύσει τον διάλογο με τα κράτη-μέλη και ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την κατεύθυνση που προτείνει η έκθεση Φιγκερέντο. Τέλος να πω ότι η Επιτροπή θα ενθαρρύνει την, τις διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου για τις πρωτοβουλίες που θα αναλαβούν, τόσο ώστε να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις, τη στρατηγική αυτή. Και θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα λάβει θέση για να υποστηρίξει τους στόχους που υποβάλλονται για την νέα ισότητα ανδρών γυναικών. Δεν θέλω να σχολιάσω τα διάφορα σημεία που θα οδηγήσουν σε που θα μπουν στην ουσία των συζητήσεων είναι πρόημα νομίζω. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να λάβω θέση. Ευχαριστώ κύριε Φίνα. Για να κλείσει η συζήτηση θα δώσω ξανά το λόγο στην κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν το λόγο και συνεργάστηκαν στην προετοιμασία του κειμένου. Βοήθησα νομίζω την βελτίωση της ποιότητας της έκθεσης. Ευχαριστώ όλους και για τις προτάσεις που υπέβαλαν και θα τους ζητούσα να μου στείλουν γραπτό τι ε, τροπολογίες τους μέχρι τις 9 αν δεν κάνω λάθος που είναι η τελική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Θα έλεγα λοιπόν όποια τροπολογία έχετε ή θεωρείτε σκόπιμη μπορείτε να την υποβάλλετε. αν θέλετε να υποβάλλετε νέες προτάσεις ή να αλλάξετε τις εφιστάμενες, λαμβάνοντα υπόψη και αυτά που σας παρουσίασα, με χαρά να σας δω. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλα τα ζητήματα. Και να μπούμε διεξοδικότερα ίσως σε κάποιες πτυχές του θέματος. Υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ που, θέλω, που το υπογράμμισαν κάποιοι συνάδελφοι. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική βούληση από πλευράς όλων. Συμβουλίου Επιτροπής και των μελών και Κοινοβουλίου προφανώς. Για να προχωρήσουν ουσιαστικά και πρακτικά τη στρατηγική για την ισότητα. Προφανώς μπορούμε να γράψουμε τα ωραιότερα κείμενα του κόσμου χάρτη, θε να τον πει, στρατηγική θε να τον πει. Ωραία και καλά είναι όλα αυτά. Όμω, αν την επαύριο η πλειοψηφία ξεχνάει το τι έχει γράψει, δεν κάνουμε τίποτα. Και αν δεν υπάρχει πρακτική συνέχιση των αποφάσεων, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γι' αυτό στην έκθεση προσπάθησα να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα της πολιτικής ε, παρέμβασης και την ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν όλοι, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, ως προς την ανάγκη να υπάρξουν κάποια νέα πολιτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την υλοποίηση αυτής της μόνιμης παρακολούθησης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι σημαντική αυτή η ετήσια συνάντηση με τους διέφερους εμπλεκόμενους για να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Γι' αυτό θέλω να υπάρξει μια μεγάλη ετήσια σύνοδος με παρουσία γυναικών, με παρουσία συνδικάτων και με ευαισθητοποίηση των κρατών μελών, των εθνικών κυβερνήσεων, των εθνικών κοινοβουλίων γιατί αλλιώ μπορεί να φτιάχνουμε ωραίες στρατηγικές, αλλά στην πράξη να διαπιστώσουμε ότι τα προβλήματα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή της πολιτικής στρατηγικής μας και να μετατρέψουμε τη στρατηγική αυτή σε μια στρατηγική όχι μόνο τη Κομισιόν, αλλά μια στρατηγική όλων, ιδίω δε του Συμβουλίου του ίδιου. Αυτό, αυτά θα ήταν τα σημαντικά πολιτικά βήματα για να υπάρξει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή τη ε, μάχη για την ισότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να μείνουμε μόνο σε θεωρητικές μενίες, αλλά να αναζητήσουμε τα σωστά πρακτικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να υπάρξει μια ετήσια παρακολούθηση της εξέλιξης και θα επιτρέψει την αλλαγή της κατάστασης. Ευχαριστώ όλους και όλες. Περιμένω τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φιγκέρδο. Προθεσμίες. Τροπολογίες. Τελευταία προθεσμία 9 Απριλίου 12. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 3-4 Μαΐου και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Τελειώσαμε το σημείο 6. Προχωρούμε στο σημείο 7 που αφορά την πορεία προς το 2014, τις σχέσεις μεταξύ γυναικών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για τη συμπεριφορά των γυναικών στις ευρωεκλογέ με παρουσίαση από την κυρία Κράτσα, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής μας. Κυρία Κράτσα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με προοπτική το 2014. Πήρα αυτή την πρωτοβουλία να ζητήσω να εντάξουν αυτό το θέμα, διότι ε, τον Μάρτιο, στις 2 Μαρτίου, με την ευκαιρία της ε, Παγκόσμιας ημέρας για τις γυναίκες, ε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, είχαμε ένα σεμινάριο με αυτό το θέμα ακριβώς. Ορίζοντας 2014 ποιες οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γυναίκες. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της συζήτησης και είχε πολύ πενιχρή συμμετοχή των μελών της Επιτροπής μας. Έτσι αποφάσισα να προτείνω να ξαναφέρουμε το θέμα αυτό της συζήτησης διότι ε, έχει να κάνει ευρύτερα με μια Ευρώπη ζωντανή, με μια Ευρώπη κοντά στις γυναίκες όπως θέλουμε εμείς να την υπηρετήσουμε και όπως βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε να φτάσουμε αυτό το στόχο. Ε, το, σεμινάριο αυτό ήταν βασισμένο στα αποτελέσματα ερευνών που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών ε, του περασμένου Ιουνίου. Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για να καταστρώσουμε τη στρατηγική μας για τις επόμενες εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικά και για το καθημερινό μας έργο. Να γνωρίσουμε δηλαδή ποιες είναι οι επιδιώξεις των γυναικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πού εμείς μπορούμε να ανταποκριθούμε, ποια είναι η άποψη που έχουν οι γυναίκες, πώς μπορούμε αυτή την άποψη όπου είναι σφαλμένη να τη διορθώσουμε και πώς θα αξιοποιήσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτουμε για αυτό το στόχο. Καταρχάς θέλω να σας πω η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο από τους άνδρες αποστασιοποιημένες από την Ευρωπαϊκή ε, ε, από, την, το χτίσιμο της Ευρώπης και από την διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας που είμαστε γυναίκες πολιτικοί δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό μοιραίο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, αδράξουμε κάθε ευκαιρία, να αξιοποιήσουμε κάθε μέσο για να αλλάξουμε αυτό, αυτή τη σχέση. Και πρέπει να δούμε τι μπορεί να παίξουμε, ε, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο τι μπορούμε να κάνουμε παράλληλα εμείς η κάθε μια γυναίκα, οι γυναίκες με τη δέσμευση που έχουμε, γυναίκες πολιτικοί, τι μπορεί να κάνουν οι πολιτικές μας ομάδες, τι μπορεί να κάνουν τα πολιτικά μας κόμματα στην πατρίδα μας. Πολλές φορές έχουμε θέσει αυτές τις προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σοβαρά εν ώψη του 2004 αν θέλουμε να έχουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή μεγαλύτερη ανταπόκριση στις εκλογές του 2014. Καταρχάς αυτό στον πυρήνα του προβληματισμού μας είναι ένας σάχλε θα έλεγα στα γαλλικά, ε, ένας φαύλος κύκλος ε, στη σχέση μεταξύ γυναίκε, γυναίκες και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν, δεν διαισθάνονται, δεν αντιλαμβάνονται τη συνέπεια, την επίδραση που έχει η ευρωπαϊκή πολιτική στη ζωή τους. Αφού δεν καταλαβαίνουν αυτή την επίδραση, είναι αποστασιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αισθάνονται ότι είναι κάτι που δεν τις αφορά. Όσο αποστασιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο λιγότερες ευκαιρίες έχουν να ενημερωθούν για αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ζωή τους και το μέλλον τους και να επιδράσουν με τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ακόμη περισσότερο κοντά τους. Λοιπόν, εμείς έχουμε ε, μια μεγάλη πρόκληση ε, απέναντί μας να αντιμετωπίσουμε αυτό τον cercle vicieux που υπάρχει στη σχέση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και γυναίκες. Εδώ η Επιτροπή μας έχει δώσει μάχες με αποτελέσματα κρατάει ζωντανή τη φλόγα της, ε, του προβληματισμού, της ανάλυσης, των πολιτικών παρενέσεων και των πολιτικών αποφάσεων όπου έχει ένα αποφασιστικό ρόλο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύτερα θα έρθουμε πιο κοντά στις γυναίκες ε, κάνοντας, ε, δίνοντας μεγαλύτερες ε, εξηγήσεις και προσεγγίζοντας περισσότερο όσον αφορά το έργο μας. Από τα αποτελέσματα των ερευνών φαίνεται ότι στον πυρήνα του έργου μας πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Δεν είναι κάτι καινούριο που πρέπει να πούμε στην Επιτροπή μας και οι συζητήσεις που προηγήθηκαν και οι συζητήσεις που έπονται έχουν να κάνουν με τις ανισότητες που ακόμη υπάρχουν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή. Βασικά, οι ανισότητες στους μισθούς. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι 50% ε, περίπου των Ευρωπαίων αντιλαμβάνονται αυτή την ανισότητα. 52% είναι στις γυναίκες, 48% είναι στους άνδρες μία μεγαλύτερη προσπάθεια αν κάνουν οι άνδρες. Και εμείς για να εξηγήσουμε στους άνδρες θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ένα ισόρροπο αποτέλεσμα στην ε, ε, συνειδητοποίηση αυτού του προβλήματος. Ε, είναι κάτι το φέρνω ως παράδειγμα, διότι βρίσκεται στον πυρήνα της ανισότητας, αλλά είναι και κάτι στο οποίο η Επιτροπή μας δίνει μεγάλη σημασία. Τονίστηκε, θα ξανατονιστεί και μπορούμε να δούμε πώς εμείς μπορούμε να λάβουμε μια δράση πολιτική που να αφήσει ένα μήνυμα αυτού του προβληματισμού και αυτού του στόχου που είναι η αντιμετώπιση της ανισότητας, πώς μέσα από, το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Μπορούμε να στείλουμε ε, μηνύματα ε, ε, σε όλη την επικράτεια, χρησιμοποιώντας τα διαδραστικά μέσα που έχει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη Web ε, τα, τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία μετέχει το Κοινοβούλιο, μπορεί κάλλιστα μια στοχευμένη δράση της Επιτροπής μας να ε, δημιουργήσει ένα θέμα συζήτησης, θέμα προβληματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διπλό στόχο. Την ευαισθητοποίηση για την ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της διάκρισης, αλλά θα στείλει ένα μήνυμα το πόσο απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιο μπορεί να φανταστεί ότι ένα μεγάλο μέρο των συζητήσεών μα σήμερα ε, και του πάθους που εκφράζουμε. Ε, είμαι σίγουρη ότι και στην επόμενη έκθεση συζήτησης θα έχουμε το ίδιο θέμα προς αντιμετώπιση. Έχουν να κάνουν αυτό το θέμα. Λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε τα μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πέρα από τα άλλα μέσα που έχουμε εμείς ως πολιτικοί, οι πολιτικές μας ομάδες, για να στείλουμε αυτό το μήνυμα της έννοιας μας, της παρένεσης και του στόχου που έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Άλλο θέμα είναι το θέμα της εναρμόνισης των οικογενειακών και βαρών και των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα σας έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος, ε, ε, κοντά στο 70, είναι 79% των γυναικών, 72% των ανδρών, αναγνωρίζουν την επιβάρυνση αυτή των γυναικών. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή συμμάχους και εταίρους στην καμπάνια, στην εκστρατεία που θα κάνουμε το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Μένει όμως να κάνουμε γνωστά αυτά τα οποία εμείς κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να εντάξουμε σε όλες τις πολιτικές ε, και σε όλες τις αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Άλλο θέμα είναι ε, το... Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι αν περάσουμε το μήνυμα ότι έχουμε συνέσεις των διακρίσεων. Και είναι η αιχμή του δόρατος στο αγώνα μας η αντιμετώπιση των διακρίσεων, οι γυναίκες οι οποίες είναι αποστασιοποιημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πιστεύουν ότι δεν ασχολείται με τα προσωπικά τα καθημερινά προβλήματα, θα αλλάξουν εικόνα. Άλλο στόχος μας πρέπει να είναι η, η ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά και ο αγώνας που κάνουμε για να το πετύχουμε και εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα. Ε, δεν είναι μόνο στα πολιτικά κόμματα, είναι στις επιχειρήσεις. Ε, μια έκθεση την οποία θα έχουμε ε, στη συνέχεια έχει να κάνει με το θέμα αυτό, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχυθεί η γυναικεία παρουσία στα κέντρα των αποφάσεων στις επιχειρήσεις. Δεν αρκεί να μείνουμε μόνο θαυμάζοντας την Ορβηγία. Πρέπει να δούμε πώς εμείς έχουμε καλές πρακτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε, όπως πρόσφατα είναι το παράδειγμα της Γαλλίας που παίρνει ε, αυτές τις ε, νομοθεσίες, τη σχετική νομοθεσία. Ε, το άλλο θέμα είναι ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική που, παρέμβαση σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο εθνικό λιγότερο, σε επίπεδο ευρωπαϊκό ακόμη λιγότερο. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε σαφές ότι η ευρωπαϊκή πολιτική είναι μια πολιτική ανθρώπινη, είναι μια πολιτική ανθρωποκεντρική, είναι μια πολιτική που έχει ε, ε, οριζόντια στόχο του την ε, αντιμετώπιση των διακρίσεων και την προώθηση του ρόλου και των ευκαιριών στις γυναίκες, διότι πράγματι είναι στις αξίες και στους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, αυτή η, η οριζόντια διάσταση, το gender mainstreaming και ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει γυναικείο πρόσωπο, διότι είμαστε ένα ποσοστό γυναικών πάνω από το εκπροσώπων γυναικών πάνω από το 1 τρίτο και ένα ποσοστό πολύ, ε, αρκετά αισθητά μεγαλύτερο από ότι είναι σε, ε, στα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μπορούμε να το κάνουμε προς τα έξω περισσότερο γνωστό, ε, κάνοντας έτσι δελεαστικό το ο, το θεσμικό μας όργανο ε, και πιο με μεγαλύτερη εκτίμηση, δίνουμε μεγαλύτερη εκτίμηση και προσοχή στην πολιτική μας. Και επειδή αυτά για να, για να χτίσουμε ένα νέο πρόσωπο, για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ε, γυναίκες, ε, ε, χρειάζεται χρόνος. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτά τα πολύτιμα αποτελέσματα της έρευνας που έχουμε, που με λεπτομέρειες τις έχετε στο φάκελό σας, μπορείτε να, να τα βρείτε, να τα επεξεργαστείτε, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία, που έχουν κάνουν με γενικά συμπεράσματα, αλλά και με, με ειδικά συμπεράσματα για κάθε χώρα ε, θα είναι πολύτιμα εργαλεία για την καθημερινή μας δουλειά, για την κάθε μια από εμά, τον κάθε ένα από εμά, αλλά θα είναι και τα εργαλεία πάνω και τα δεδομένα πάνω στα οποία θα καταστρώσουμε τη στρατηγική μας για τις επόμενες ευρωεκλογές. Στόχος μας είναι όσο τα δω περισσότερες γυναίκες στις κάλπες, χωρίς να αποτελούν ένα ειδικό στόχο οι γυναίκες, διότι μέσω όρο έχουν δύο μονάδες διαφορά λιγότερο ψηφίζουν, ποσοστό γυναικών που ψηφίζουν από ότι οι άνδρες. Υπάρχουν δε και κάποιες χώρες που οι γυναίκες ψηφίσαν περισσότερο και από τους άνδρες. Άρα από, στόχο ιδιαίτερα δεν αποτελούν οι γυναίκες να τι ε, να ε, κάνουμε να πάνε στις κάλπες. Στόχος μας είναι να μας προσέξουν για να αισθανθούν ότι είναι η Ένωση μια Ένωση ε, ανθρώπινη, μια Ένωση που υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, που υπηρετεί τις ίσες ευκαιρίες είναι πραγματικά ε, ένα πολιτικό σχέδιο πολύ κοντά στις γυναίκες. Και χρειαζόμαστε την προσοχή των γυναικών, όχι μόνο για να μας ανταμείψουν στις εκλογές, αλλά όσο αισθάνονται ότι είμαστε μακριά από αυτές, τόσο λιγότερο ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας και να συνδιαμορφώσουν την Ευρώπη του αύριο. Ήθελα να σας πω ότι οι υπηρεσίες ε, επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στη διάθεσή σας. Ε, τόσο οι υπηρεσίες του press service όσο και οι υπηρεσίες των μελετών και της επεξεργασίας των δεδομένων ε, και θα είναι μια ευκαιρία για μένα, καταλαβαίνετε, ως αρμόδια αντιπρόεδρο για την επικοινωνία και μέλος πιστό της Επιτροπής ε, επί 10 χρόνια, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο συνδυασμό, ούτω ώστε και το έργο της Επιτροπής μας να φανεί και την υπόθεση των γυναικών να υπηρετήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κράτσα για όσα μας είπατε. Ήταν μια πολύ εμπεριστατωμένη εισαγωγή σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αυτή την πάρα πολύ σημαντική μελέτη την οποία θα πρέπει να αναλύσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και να τη σκεφτούμε όλοι μας για να συναγάγουμε κάποια νέα συμπαράσματα και να έχουμε νέες ιδέες για τις επόμενες εκλογές. Είχα το προνόμιο να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ των μελών και των εμπειρογνωμόνων που ανέλησαν την μελέτη και αναλύουν τη μελέτη και, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες και κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή τη συνάντηση. Πιο συγκεκριμένα προβληματίζομαι όσον αφορά την στάση των γυναικών ε, έναντι των εκλογών. Η αντιπρόεδρός μας τα είπε πολύ ξεκαθά τα πράγματα πιστεύω. Υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη ενδιαφέροντος στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες όσον αφορά τις ευρωεκλογές. Και αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη πληροφοριών. Και γι' αυτό οι γυναίκες δεν κατανοούν γιατί οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι τόσο σημαντικές. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή και δεν καταλαβαίνουν πώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζουν και τις εθνικές πολιτικές. Ούτε αυτό το κατανοούν. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε ε, πώς οι γυναίκες πηγαίνουν να ψηφίσουν υπάρχει ε, μικρότερη αποχή όταν στον εκλογικό κατάλογο υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Μπορούμε κάτι να μάθουμε από αυτό. Αυτό ισχύει περισσότερο στις σκανδιναβικές χώρες. Επίσης είναι σημαντικό να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τις γυναίκες υποψήφιες. Ε, είναι, είναι λιγότερο ορατές στα μέσα ενημέρωσης οι γυναίκες όταν είναι υποψήφιες. Προβάλλονται λιγότερο. Και όταν προβάλλονται στα μέσα ε, δεν προβάλλονται για τους σωστούς λόγους πάντα. Ο τρόπος με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι γυναίκες υποψήφιοι είναι διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τα μέσα ενημέρωσης οι άντρες υποψήφιοι στην Πορτογαλία καλύπτονται οι γυναίκες ε, στα μέσα ενημέρωσης λόγω εμφάνισης, λόγω του τρόπου ενδυμασίας τους, λόγω της γενικής εικόνας που προβάλλουν, λόγω της οικογένειάς τους ή ίσως λόγω εργασίας συζύγου. Αλλά δεν προβάλλονται λόγω πανεπιστημιακών ιδιωτήτων, ε, λόγω του επαγγέλματό τους ή της πολιτικής δουλειάς που κάνουν. Ενώ οι άντρες προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης λόγω του βιογραφικού τους, λόγω τη παρελθούσα δουλειά τους, της παλιά τους πολιτικής θέση κλπ. Και το καθεξής. Τα μέσα ενημέρωσης λοιπόν αναπαράγουν τα κοινωνικά στερεότυπα όσον αφορά τους ε, άντρες και τις γυναίκες. Τα μέσα ενημέρωσης δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν ε, σαν σοβαρούς ανθρώπους τις γυναίκες, τις προεκλογικές ε, περιόδους. σαν αναξιόπιστους ανθρώπους. Η χρήση όλων των μορφών μέσων ενημέρωσης και των μίντια κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουν καλύτερα οι γυναίκε υποψήφοι. Να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα μέσα ενημέρωση οι γυναίκε υποψήφοι. Πολλέ ήταν επιτυχεί χρησιμοποιώντα το διαδίκτυο και άλλα δίκτυα για να περάσουν το μήνυμά του. Να περάσουν σοβαρά μηνύματα είδαμε κάποιες γυναίκες που βελτίωναν την αξιοπιστία τους και την, ε, το συνέστημα ότι είναι ικανές χρησιμοποιώντα τα κοινωνικά αυτά δίκτυα, την κοινωνική δικτύωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να συνεχίσουμε τη συζήτηση στο μέλλον, είναι σημαντικό να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, τόσο ώστε το 2014 οι γυναίκες υποψήφιες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπιστούν πιο ισότιμα στα μέσα ενημέρωσης. Η κυρία Οβίρ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εφόσον εσείς τελειώσετε αναφέροντας τα ΜΜΕ, θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω με αυτά, παρά το ότι βεβαίως τα ΜΜΕ είναι ένα δεύτερο επίπεδο που χαρακτηρίζει τις γυναίκες με βάση το ότι αυτές φοράνε. Στην Εστονία πριν από λίγα χρόνια ανέλησαν τα σχολικά βιβλία και βλέπουμε και σε άλλα κράτη-μέλη πως τα σχολικά βιβλία ε, υπάρχει μια μητέρα που φοράει ποδιά και ο πατέρας στέκεται δίπλα στο αυτοκίνητο. Διάβασα εγώ αυτά τα έγγραφα λοιπόν πολύ προσεκτικά την ανάλυση αυτή και για να είμαι ειλικρινής για πρώτη φορά έλαβα αυτό το υλικό εγκαίρος γιατί έχουμε καιρό μέχρι τις ε, επόμενες εκλογές. Βεβαίως οι γυναίκες είναι παγιδευμένες σε ένα φαύλο κύκλο, δεν θεωρούν ότι μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικό ρόλο στις ζωές τους. Αυτό σχετίζεται και με το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Οι γυναίκες θέλουν αποτελέσματα, λιγότερη φτώχεια, περισσότερη δουλειά, ίση αμοιβή. Και τα έχουμε συζητήσει αυτά τα πράγματα εδώ εδώ και πολύ καιρό. Ακόμα και τα ΜΜΕ δεν μας δίνουν πια σημασία και δεν καλύπτουν ούτως ή άλλως το τι λένε οι γυναίκες. Και παραδείγματο χάρη στην περίπτωσή μου μου λένε «Μα μόλις σας πήραμε συνέντευξη» ενώ ήταν πριν από δύο ολόκληρους μήνες. Οπότε πρέπει να είμαστε πιο ισχυρές, συνεπείς και να εγγυηθούμε πως οι αποφάσεις μας ε, θα τηρούνται και θα έχουν αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο ίσως ε, μπορέσουμε ε, να επιτύχουμε το να θεωρούν οι γυναίκες πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ζωή τους. Όπως είπα, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό επίβλεψης και εφαρμογής για να εφαρμόζει τις αποφάσεις μας. Από την άλλη, δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως ο μισός πληθυσμός της Ένωσης είναι γυναίκες. Και αν εξακολουθούν να θεωρούν πως δεν είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βλέπουν τα αποτελέσματα του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κάνουμε, διαλύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξακολουθεί βέβαια ο κόσμος να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ο κίνδυνος, ε, τα πιο ακραία στοιχεία να εκλεγούν εδώ πέρα και δεν νομίζω πως ε, είναι σωστό κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο 7 και να πάμε στο σημείο 8. Η έκθεση Ρωμέβα Ιρουέδα για τις πτυχές ισότητας των φύλων όσον αφορά την οικονομική ύφεση και χρηματοστατικής κρίσης. Έχουμε 144 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. ο εισηγητής έχει δουλειά μπροστά του. Αν θέλει να καταλήξει σε κάποιες συμβιβαστικέ ε, λύσεις στο εγγύς μέλλον. Ο κύριος Ρωμέβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα να μιλήσω και στο προηγούμενο σημείο γιατί νομίζω ότι σχετίζονται. Ακριβώς η αντίληψη που αναφέρει η έκθεση του ότι τα πολιτικά θέματα στην Ευρώπη επηρεάζουν λιγότερο ή δεν επηρεάζουν ή επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες είναι σημαντική για να καταλάβουμε το πώς συνδέεται η συζήτηση αυτή με την έμφαση που δίνουμε στις κρίσεις, την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική, την κοινωνική που βιώνουμε. Συνδέονται τα θέματα αυτά και σε ό,τι αφορά και σε σχέση με την ανάλυση του Ευρωβαρομέτρου και σε σχέση με την έκθεση αυτή, γιατί σημαίνει έκθεση λέμε τι θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να καλύψουμε το κενό αυτό, να εξηγήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο ποια είναι όχι μόνο τα προβλήματα που επηρεάζουν τις γυναίκες από την οπτική, από την έμφυλη διάσταση, αλλά κυρίως ποιες είναι οι προτάσεις με ευρωπαϊκό όραμα που θα βοηθήσουν να σπάσει αυτή η δυναμική, η απομόνωση, η απευθείας περιθωριοποίηση. Συνδέονται λοιπόν τα δύο πράγματα. Είναι γεγονός ότι η έκθεση δημιούργησε ένα κάποιο ενδιαφέρον, 140 τόσες τροπολογίες, τέλος τέλος. Είναι μάλλον ψηλός αριθμός τροπολογιών. Πολλές, ωστόσο, τροπολογίες προτάθηκαν δεν θα υπάρξουν δυσκολίες από πλευράς μου να δεχθώ τις, τη μεγάλη πλειοψηφία τους. Είναι ενδιαφέρον το ότι υπάρχει μια συνένεση, μια σύμπτωση απόψεων από όλες τις πολιτικές ομάδες ως προς την ανάγκη να υπάρξουν στοιχεία που θα εμπλουτίσουν το κείμενο. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά τροπολογιών που υπέβαλαν πολλές συνάδελφοι που είναι, αποτελούν προσθήκη, δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Τις δέχομαι τις περισσότερες. Κάποιες άλλες θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο συμβαστικής λύσης, διότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ιδεολογικού χαρακτήρα. Π.χ. Ο, λόγο, ρόλος των ε, δημοσίων υπηρεσιών, η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια, ο ρόλος των γυναικών σε όταν αφορά την πρόσβαση, την πρόσβαση σε κάποιες ε, ε, σε κάποιους τομείς δυνατοτήτων τους. Εγώ θα προσπαθήσω να υποβάλω κάποιες προτάσεις συμβιβαστικού χαρακτήρα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχουν τροπολογίες, αρκετές τροπολογίες, και αυτό με εξέπληξε, όπου υπάρχει πρόθεση να φύγουν τμήματα του κειμένου. Κάποιες από αυτές, γι' αυτό μιλούσα για την προηγούμενη έκθεση, στην πράξη καταργούν στοιχεία που σχετίζονται όχι με θέσεις αλλά με δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, παραπομπές σε συγκεκριμένα κείμενα της Επιτροπής, παραπομπές σε συγκεκριμένα κείμενα, σε συγκεκριμένες μελέτες να σας πω την αλήθεια, αυτό με έχει εκπλήξει λίγο, με έχει ανησυχήσει. Γιατί βλέπω ότι κάποιες τροπολογίες θέλουν να βγάλουν από το κείμενο στοιχεία που θεωρώ κρίσιμα, όχι μόνο για να έχουμε μια εικόνα του πλαισίου, αλλά για να αποδείξουμε σαφώς ότι η Επιτροπή έχει να πει κάτι θετικό Αυτές είναι τροπολογίες που προέρχονται κυρίως από, ένα, από μια πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ. Θα προσπαθήσω λοιπόν σε διμερές επίπεδο να δω κατά πόσον υπάρχει πραγματική βούληση κατάργηση κειμένου ή μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμβαστική λύση. Θα έλεγα λοιπόν ότι είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι υπάρχει μια συνένεση ως προς την ύπαρξη του προβλήματος, στο ότι τμήμα της λύσης μπορεί να προέλθει από πλευράς Ένωσης και μια συνένεση για το ότι η Επιτροπή μας μπορεί να προσφέρει κάτι χρήσιμο. Αυτό είναι η αφετηρία και ελπίζω και το και ο τερματικό σταθμό της έκθεση μου. Έχω ένα χρονοδιάγραμμα. 14 Απριλίου για να κλείσουμε τις συμβαστικές προτάσεις και ελπίζω μέχρι τότε να έχω ετοιμάσει το κείμενο και να ξεκινήσω τη διαπραγματεύση. Ευχαριστώ. Κύριε Δομέβα, η κυρία Κλάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο μόλις είπατε. Πρώτα απ' όλα το θέμα αυτό των πτυχών των φύλων στην οικονομική ύφεση και την κρίση. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε στις λεπτομέρειές του και πράγματι αυτό κάνατε, το κάνατε πολύ καλά, κατά την άποψή μου με έναν τρόπο ο οποίο βεβαίω μπορεί να γίνει. Πράγματι μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα εάν θέλουμε μόνο να δούμε πόσο επηρεάζονται οι γυναίκες βεβαίως μπορούν ε, να επηρεαστούν αρνητικά εξίσου και οι άντρε Γι' αυτό εγώ έχω κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα με αυτή την έκθεση. Δυσκολεύομαι κάπως γιατί τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτά τα οποία έχουμε βάλει σε όλες μα όλες τις εκθέσεις ε, τα βάζουμε και εδώ πέρα με άλλο τίτλο σχετικές δηλαδή με την ισότητα των φύλων, πτυχές οικονομική ύφεση και τη χρηματοπιστωτική κρίσης. Όποια έκθεση και να γράψουμε δηλαδή, σε ένα συνολικό πλαίσιο, ε, έχουμε ένα πρόβλημα. Αν το δούμε μόνο στο ζήτημα της οικονομικής ύφεση και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που είναι ο τίτλος βεβαίως, τότε πρέπει να είναι πιο στενότερο μικρότερο και ουσιαστικότερο το κείμενο. Εξού και οι τροπολογίες που έχω κάνει που είναι προτάσεις διαγραφής. Δεν είναι τώρα δουλειά μας εδώ πέρα να μιλήσουμε για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. και βλέπουμε εδώ πέρα και τις διαφορές ε, που έχουμε μεταξύ των κομμάτων. Αν δείτε π.χ. το σημείο 14 αναφέρεται πράγματα τα οποία είναι ε, πράγματα ε, αδιαμητρότητας και τα οποία αφενός είναι ρευστά, δεν έχουν σχέση εδώ πέρα με το θέμα μας. Σημείο 15. Οι εθνικοί νόμοι να βελτιωθούν όσον αφορά τη βία των Τι σχέση έχει αυτό με την χρηματοπιστωτική κρίση. Ή, εντάξει, εδώ μπορεί να διαφωνήσουμε τέλο πάντων σε αυτό. Που λέτε οι άντρες και οι γυναίκες ε, να έχουν θέσεις, ε, ε, να εκπροσωπούνται εξίσου στις θέσεις αποφάσεων. Ξανά και ξανά τις ίδιες απαιτήσει έχουμε, αλλά αυτά δεν αφορούν ειδικά την κρίση. μιλάτε μετά για το ποσοστό γυναικών που πρέπει να ανέβει στο 40% στις ανώνυμες εταιρείες και τα δουσού. Και μετά σημείο 19, πράσινη τεχνολογία και εξυγχρονισμός των υποδομών. Τα πάντα δηλαδή έχετε βάλει εδώ πέρα. Ε, εντάξει, παραπάει λίγο, είναι, παρά είναι λίγο βαρύ και είναι γύρω γύρω από το θέμα, δεν έχετε αγγίξει το θέμα. Ξέρω πως είναι δύσκολο θέμα, αλλά ε, πρέπει να το ξαναδείτε από την αρχή. Οι 144 τροπολογίε κάτι πρέπει να σας πούν. Ότι πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν έρθει βεβαίω τώρα τέτοια ώρα εδώ πέρα αλλά διαφωνούν και δεν συμφωνούν με την προσέγγιση που έχετε εδώ πέρα στο θέμα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, κάνατε πολλή δουλειά, αλλά το, το θέμα, δεν ξέρω, το έχετε προσπεράσει. Δεν ξέρω, ειλικρινά και αν ε, βοηθάμε τις γυναίκες έτσι. Οποιοδήποτε πρόβλημα στον κόσμο μετά να πούμε έχει και μια πτυχή γυναικεία. Ε, δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει και... Το λέτε κιόλα, δεν υπάρχει στρατιστική ε, που να αναφέρει ειδικά την επίδραση της κρίσης για τις γυναίκες. Οπότε έχω πρόβλημα εγώ αρχής και με το θέμα και με αυτά τα οποία τελικά καταλήξατε να γράψετε. Οπότε σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω εγώ ως σκιώδης εισηγήτρια για την ομάδα μου. Για να πω και εγώ δύο πράγματα. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν 144 τροπολογίες. Όντως, αυτό όμως είναι δείγμα της σπουδαιότητας του θέματος αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι κάποιες τροπολογίες ε, έγιναν δεκτές χτες μόνο. Σε δύσκολες γλώσσες κάποιες από αυτές, για μένα τουλάχιστον ελληνικά, γερμανικά, ούτε και τα πορτογαλικά δηλαδή είναι εύκολη, συνηθισμένη γλώσσα, εκτός από μένα. Και αυτό δυσχεραίνει την αξιολόγηση όλων των υποβληθήσεων προτάσεων. Όμως, μετά από μια πρώτη ανάγνωση, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη μεγάλη δουλειά που έκανε ο εισηγητής. Προς την κατεύθυνση αυτή πηγαίνουν και οι τροπολογίες μου άλλωστε. Να αναδείξουμε τη συμβολή των γυναικών στην έξοδο από την κρίση. Να υπογραμμίσουμε ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο υπεύθυνε για την προέλευση και τις αιτίες της κρίσης. Και αυτό είναι κάτι Ούτε μία γυναίκα δεν υπάρχει διοικητής κεντρικής τράπεζας στα 27 κράτη-μέλη. 5% των γυναικών, 5% μόλον, μάλλον των ε, ε, ηγετών, των ηγετικών θέσεων στα μεγάλα, στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι γυναίκες. Η μη παρουσία λοιπόν γυναίκας στα όργανα αυτά δείχνει ότι δεν ήταν οι γυναίκες υπεύθυνε. Για καλό για κακό, αυτές που προκάλεσαν ή που θα μπορούσαν να προλάβουν την κρίση. Αλλά οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα της κρίσης. Και η έμφυλη βία έχει ε, παίζει, και, και στην έμφυλη e βία παίζει ρόλο η κρίση. Έχουμε πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που δείχνουν ότι αυξήθηκε η βία μετά την κρίση και ως συνέπεια της κρίσης. Η αύξηση της ανεργίας, η, η υπερχρέωση της οικογένειας, η αύξηση της, ε, των δυσκολιών, η έλλειψη εσόδων δημιουργούν με τη σειρά τους επιθετικότητα, αστάθεια στον οικοκυριό την αιστεία και τα θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Σας ευχαριστώ επίσης την προσοχή του εξή. Εγώ μετλέτησα το θέμα αυτό και ε, είχα μετάσχει σε μια συνάντηση στη χώρα μου όπου μίλησα για να προσπαθήσω να... Και για να μιλήσω αυτή την ομιλία είδα μια σειρά μελετών μεταξύ των οποίων μιας υπηρεσίας ε, μια, ενός μιας βρετανικής εταιρείας που δείχνει ότι επιχειρήσεις στις οποίες στα, δι, ε, που έχουν διοικητικά συμβούλια με ε, παρουσία γυναικών τουλάχιστον τριών τον αριθμό, που είναι το απαραίτητο μήνυμο για να επηρεάσουν στη λήψη της απόφασης, αποδείχθηκε ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις πήγαν καλύτερα στο χρηματιστήριο σε 83% των περιπτώσεων και έδωσαν, έφεραν δηλαδή κέρδη λόγω ανάπτυξης, λόγω αποτελε, οικονομικών αποτελεσμάτων αυξημένα κατά έως και 73%. Δηλαδή οι γυναίκες μπόρεσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους. Όταν σε διοικητικά συμβούλια, μάλλον επιχειρήσεις με διοικητικά συμβούλια στα οποία υπάρχουν τουλάχιστον τρεις γυναίκες. Στην οδηγία, για παράδειγμα, μια συντηρητική κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία να θέσει ποσόστοση παρουσίας των γυναικών στις δημόσιες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που το ακολουθεί και η Γαλλία. Αλλά, αλλά τι σημαίνει αυτό. Για οικονομικούς και μονολόγους πρέπει να θεωρήσουμε πλεονεκτικό το να αυξήσουμε την παρουσία των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις και την εργασία του εισηγητή και με πολλές από τις προτάσεις που, που έχουν υποβληθεί που σίγουρα θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε συμφωνίες και να επιστήσουμε την προσοχή στην σπουδαιότητα που παίζουν οι γυναίκες στην οικονομική δραστηριότητα. Όχι την πολιτική μόνο. Εδώ και καιρό λέμε κάτι τέτοιο. Τελειώνω. Είμαι έτοιμη να προχωρήσω σε συμφωνίες για να επιτύχουμε μια συνένεση και να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση, γιατί πιστεύω ότι είναι μια σημαντικότατη έκθεση και εξαιρετικά επίκαιρη. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θέλει και η Κομισιόν να μετάσχει στη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Οζάν έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης ε, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε πόσο ενδιαφέρον και χρήσιμο είναι να ξέρουμε τις συνέπειες της κρίσης για τις γυναίκες. Κάτι που καλύψαμε σε πολλά κείμενα της Επιτροπής, την κοινή έκθεση για την απασχόληση ιδίω, την πρόσφατη έκθεση για την ισότητα των γυναικών του 2010 και την ανάλυση του αντίκτυπου της κρίσης στην αγορά εργασία. Και θα καταγράψουμε τα αιτήματα που θα εμφανιστούν στην έγκριση της, μετά την έγκριση της ε, τελικής έκθεσης. Ευχαριστώ. Θέλει ξανά το λόγο ο εισηγητής. Να πω ότι έχω προγραμματίσει να συναντηθώ αύριο με την Επιτροπή για να δούμε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Θα προτείνω μια σειρά συμβαστικών προτάσεων για να δούμε Πού μπορούμε να τα βρούμε εκεί που υπάρχουν διαφορές. Θα ήθελα να καταστήσω ωστόσο σαφές ότι η βασική αρχή της έκθεσης είναι η εξής. Ξεκινούμε από δύο προβλήματα. Ένα, το θέμα του φίλου ήταν απόν όχι μόνο στην ανάλυση των αιτιών της κρίσης αλλά και στις προτάσεις λύσης, τους, λύσης της. Αυτό το καταδικάσαμε πλειστάκης. Ό,τι λοιπόν δεν το λέμε εμείς στην Επιτροπή, δεν το βρίσκουμε αλλού εύκολα. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε σαν Επιτροπή. Να καταλάβουμε ότι αυτή η ειδική κατάσταση πρέπει να γίνει ορατή με τον α ή β τρόπο. Κάτι που δεν συμβαίνει αλλού. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να είναι σαφές πως ε, όντως υπάρχουν πολλά θέματα, ε, είναι εκτεταμένο το ζήτημα, αλλά ε, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Είναι το βασικό θέμα που επηρεάζει σήμερα την πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι αναγκαίο να έχουμε targets, στόχους, συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούμε να προτείνουμε, να θέσουμε, να επιβάλλουμε στην Κομισιόν στα κράτη-μέλη. συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να έχουμε και μια εικόνα των εξελίξεων. Αυτή είναι μια βασική συζήτηση στην Επιτροπή. Πολλές από τις τροπολογίες αυτό θέλουν και δεν νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα να τα συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ κύριε Ομέβα. Χρονοδιάγραμμα. Τρεις και 4 Μαΐου. ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Κλείνουμε το σημείο 8. Στα διάφορα σημείο 9. Δεν έχω τίποτα. Επόμενη συνεδρίασή μας 3 Μαΐου 3 το μεσημέρι και 4 ε, του Μαΐου 9 το πρωί. Ευχαριστώ, καλή ξεκούραση, ευχαριστώ και τους διαδμηνείς για την καλή δουλειά του. Ευχαριστώ.